Good afternoon. I would like to propose you to take your seats and start the meeting. Good. Γεια σας. Παρακαλώ καθίστε. Θα ήθελα να σας ζητήσω λοιπόν να καθίσετε για να ξεκινήσουμε χωρίς καθυστέρηση. I hate this. <laughs> Ναι, thank you very much. Good afternoon again. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε πάλι. Πριν περάσουμε στην ουσία των θεμάτων, θα ήθελα να σας ενημερώσω για δύο αλλαγές. Μία από αυτές είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία που προβλέπεται για το σημείο 7 για την έκθεση του κυρίου Κάσμαν. Αναβάλλεται για την 23η Νοεμβρίου. Και είχαμε προγραμματίσει και συνάντηση των συντονιστών σήμερα η απόφαση τροποποίησης της αντιπροσωπείας μας στη Σικελία. Οι αλλαγές όμως ε, έγιναν δεκτές μέσω γραπτής διαδικασίας, ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει συνάντηση των συντονιστών. Οπότε αν δεν ε, έχετε αντιρρήσεις μπορούμε να υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη. Άλλο ένα θέμα. Αφορά την επίσκεψη στην Ιταλία. Ξέρετε ότι η επίσκεψη αυτή προκλήθηκε από την είσοδο πολιτών τρίτων χωρών. Είχε υπάρξει μια συμφωνία για τη σύνθεση της αντιπροσωπείας. Θα επισκεφθούμε το Αγκριτζέντε, το τράπανη, τη Μίνα, το Παλέρμο, τη Λαμπεντούσα φυσικά μέχρι τις 26 Νοεμβρίου. 4 του ΕΛΚΑ, τρεις σοσιαλιστές, ένας φιλελεύθερον, ένας πράσινος, ένας συντηρητικό, ένας από την ΚΟΕ και ένας από την Ανεξάρτητη Ευρώπη. Ελπίζω να κάνετε δεκτή την πρότασή μας. Uh, ε, 2.3 It is the amendment of regulation number 810 Λοιπόν, για τον κανονισμό 810 του 2009 της 13ης ε, Ιουλίου για τον ε, κοινοτικό κώδικα για τις θεωρήσεις. Η συγητής μας ο κύριος Μισελ. Πρώτα θα ακούσουμε την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν είναι εδώ. Θα σας ζητήσω λοιπόν να παρουσιάσετε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τροποποιεί τον ισχύοντα κανονισμό. Και μετά θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Πολωνικής Προεδρίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι τιμή μου να σας παρουσιάσω σήμερα την πρώτη τροποποίηση του κώδικα για τις θεωρήσεις που εφαρμόζεται από τον Απρίλιο του 10. Μία πρώτη έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέση σε εφαρμογή του κώδικα προβλέπεται για το 2013 και θα ακολουθηθεί από τροπολογήσεις του, του κώδικα αυτού. Αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα λοιπόν δεν είναι να προκαταλάβουμε την έκθεση του 2013 δεν θεωρούμε δηλαδή ότι η σχετικά πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση δεν περιελάμβανε τις σωστές ρυθμίσεις επί της ουσίας. Ανακαλύψαμε όμως κατά τη διάρκεια της πρώτης περίοδου εφαρμογής ότι το άρθρο 3 του κώδικα που αφορά τις βίζες αεροδιαμετακόμισης περιλαμβάνει ένα λάθος και δημιουργεί προβλήματα στην εφαρμογή του δεν έχει νομική βάση ξεκάθαρη. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε λοιπόν σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στην ουσία να διορθώσουμε, να κάνουμε μια διόρθωση και αυτό δεν είναι φυσικά ε, προϊόν αξιολόγησης ε, της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής. Πέντε σελίδες είναι το κείμενο το οποίο προτείνουμε. Οφείλω να σας δώσω όμως, Πρόεδρε, κάποιες ε, εξηγήσεις για να μπορέσετε να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται με αυτή την τεχνική διόρθωση την οποία κάνουμε. Είναι ένα κείμενο το οποίο είναι δύσκολο να το διαβάσει κανείς και δύσκολο να καταλάβει την, το περιεχόμενο, την εμβέλεια της πρότασης. Να θυμίσω καταρχάς ότι έχουμε τον κανονισμό του 2001-539 που καθερώνει, καθιερώνει τις αρ, τους αρνητικούς καταλόγους και τους θετικούς καταλόγους. Αρνητικοί κατάλογοι είναι αυτοί για τους οποίους χρειάζεται βίζα για να μπει κανείς στο Σέγγεν και θετικός κατάλογος είναι αυτός που περιλαμβάνει τους πολίτες των χωρών που προέρχονται από χώρες που δεν χρειάζονται θεώρηση ουσιαστικά. Καταρχάς λοιπόν οι ταξιδιώτες που φτάνουν στις ζώνες transit των αεροδρομίων Σέγγεν και που πηγαίνουν κάπου αλλού εκτός Σέγγεν μετά, δεν έχουν ανάγκη ε, να έχουν θεωρήσεις ακόμα και αν η χώρα τους περιλαμβάνεται στον αρνητικό κατάλογο. Το Μαρόκο σαν παράδειγμα είναι στον λεγόμενο αρνητικό κατάλογο. Ο Μαροκίνος που φτάνει από την Καζαμπλάκα στο Παρίσι και συνεχίζει μετά να πάει στις Ηνωμένε Πολιτείες Εφόσον παραμένει στο αεροδρόμιο στο Παρίσι, στη διεθνή ζώνη του τράνζιτ, δεν έχει ανάγκη από θεώρηση. Αυτός ο αρνητικός κατάλογος λοιπόν δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θεωρήθηκε όμως ότι μερικές φορές για λόγους ασφαλείας ή για λόγους κινδύνου παράνομης μετανάστευσης πρέπει να επιβληθεί θεώρηση και σε πολίτες οι οποίοι περνούν μόνο από τα αεροδρόμια και μένουν στις διεθνείς ζώνες των αεροδρομίων. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουν ανάγκη από την λεγόμενη ειδική βίζα transit διαμετακόμισης αεροπορικού τύπου. Έχουμε λοιπόν εγκρίνει αυτού του τύπου την θεώρηση και έχουμε ε, προσθέσει 12 περίπου τρίτες χώρες για τους πολίτες των οποίων αυτών χωρών απαιτείται μια τέτοια θεώρηση ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούν παρά μόνο για transit. Ιράν, Ιράκ, Πακιστάν, Αφγανιστάν. Εντάσσεται λοιπόν στις θεωρήσεις και στον κώδικα των θεωρήσεων. Βέβαια υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις για τους πολίτες αυτών των χωρών. Όταν τα άτομα αυτά θεωρούνται ότι δεν αποτελούν απειλή για τη δημόσια τάξη ή όταν δεν θέτουν πρόβλημα παράνομης μετανάστευσης. Στο παρόν κείμενο σημειώνεται ότι σαν παράδειγμα οι κάτοχοι κάρτας παραμονής που έχει χορηγηθεί από τρίτες χώρες εξαιρούνται από την υποχρέωση απόκτησης ειδική βίζας αεροπορικού τύπου. Γιατί το ότι έχουν αυτή την κάρτα παραμονής ή την βίζα για μία συγκεκριμένη χώρα και αναφέρομαι στον Καναδά και στις Ηνωμένε Πολιτείε, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για να περάσουν από τα αεροδρόμια μας και μπορούν να το κάνουν αυτό χωρίς ειδική θεώρηση. Αν διαβάσετε τώρα το κείμενο του άρθρου 3, προβλέπετε μία εξαίρεση στην υποχρέωση θεώρησης αεροπορικού τύπου για αυτούς οι οποίοι έχουν βίζα ή κάρτα παραμονής από κάποιες άλλες χώρες. Χώρες του οποίου όμως τα μέσα Σέγγεν, δηλαδή που ανήκουν στο Σέγγεν, δεν καλύπτουν το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, ούτε και τη Βουλγαρία, την Ρωμανία και την Κύπρο, που δεν έχουν ακόμα θέση σε εφαρμογή το κεκτημένο Σέγγεν. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι εφόσον οι πολίτες αυτών των 12 χωρών έχουν μία κάρτα παραμονής ή μία θεώρηση η οποία έχει εκδοθεί από τη ΣΥΠΑ, μπορούν να περάσουν από τα αεροδρόμια μας χωρίς να έχουν ανάγκη αεροπορικού τύπου βίζα. Εφόσον όμως έχουν κάρτα παραμονής από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν την ανάγκη να τους χορηγηθεί η ειδική αυτή θεώρηση. Αυτό εξηγείται από το ότι η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αναφερόταν στα κράτη-μέλη τα οποία χρησιμοποιούν αυτές τις δυνατότητες, αλλά τις χώρες της Ένωσης γενικά. Αυτό καλύπτει όλες τις χώρες βέβαια, ακόμα και αυτές οι οποίες δεν ανήκουν στο Σέγγεν ή δεν είναι ακόμα μέλη του Σέγγεν χωρίς εσωτερικά σύνορα. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων λοιπόν η προσθήκη αυτή ε, εξαφανίστηκε. Εκεί που λέγαμε δηλαδή χώρες της Ένωσης χάθηκε κάπου. Το συνειδητοποιήσαμε αυτό στα πλαίσια της εφαρμογής του κώδικα και προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε το λάθος αυτό όταν επεξεργαστήκαμε το εγχειρίδιο εφαρμογής των κανόνων για την έκδοση των θεωρήσεων στα πλαίσια της εναρμονισμένης εφαρμογής του κώδικα για τις θεωρήσεις. Το εγχειρίδιο αυτό βέβαια είναι διοικητικές οδηγίες ή πρακτικές οδηγίες. Ένα τέτοιο εγχειρίδιο δεν μπορεί να αλλάξει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε νομικό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί χρήσιμο να καταθέσει τη συγκεκριμένη πρόταση η οποία διορθώνει το συγκεκριμένο λάθος το οποίο διαπράχθηκε, το οποίο δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση μια συνομοθετική ε, διάθεση. Δεν θελήσαμε εμείς να εξαιρέσουμε την Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Όχι. Απλά δεν είπαμε ότι αυτοί οι οποίοι έχουν μια βίζα από τις χώρες αυτές δεν θα πρέπει να τους επιβάλλουμε μια αεροπορικού τύπου θεώρηση είναι ένα λάθος αν θέλετε, μια παράληψη την οποία σημειώσαμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε το 2013 και την έκθεση αξιολόγησης για να κάνουμε την απαιτούμενη διόρθωση. Γι' αυτό λοιπόν καταθέτουμε την πρόταση αυτή η οποία φαίνεται περίπλοκη και τεχνική αλλά μία πρόταση η οποία σύμφωνα με την Επιτροπή είναι απαραίτητη για να διευκρινιστεί η νομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτοί οι οποίοι έχουν κάρτες παραμονής και θεωρήσεις από τις χώρες τις οποίες προανέφερα. Λοιπόν, αυτά περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη πρόταση, Πρόεδρε. Είμαστε στη διάθεσή σας για η αδίποτε ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ο κύριος Φίλιπ Γιασίνσκι από το Συμβούλιο θα λάβει τώρα τον λόγο και εν συνεχεία ο Λουί Μισελ. and gentlemen. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε. Είναι δύσκολο να πω. Συνήθω όταν απευθύνομαι στα μέλη τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, λέω από την πλευρά του Συμβουλίου. Η συγκεκριμένη πρόταση είναι τεχνικού χαρακτήρα κτλ. Εδώ σε συγκεκριμένη περίπτωση, ακόμη και με μικροσκόπιο δεν μπορεί να βρει κανείς ε, πολιτικό ε, στοιχείο πρόκειται αυτός ο κώδικας ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο το οποίο εγκρίθηκε με τη βοήθεια του Συμβουλίου στο Κοινοβούλιο και διευκολύνει την καθημερινή ζωή όσων πολιτών επιθυμούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τη ζωή των υπαλλήλων. Από ό,τι καταλαβαίνω, με την τεχνική λύση θα μπορούσαμε να, βελτιω... να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο αυτό το εργαλείο. Είχαμε δε την ευκαιρία δύο φορέ να συζητήσουμε αυτό το φάκελο στο Συμβούλιο. Τα κράτη-μέλη ουσιαστικά δεν εισήγαγαν καμία αλλαγή στο φάκελο. Δηλαδή, ε, τους ικανοποίησε ε, αυτό που έλαβαν από την Κομισιόν και φαντάζομαι τις επόμενες δύο ημέρες ε, σε επίπεδο κορεπέρ θα εγκριθεί επισήμως αυτό το έγγραφο. Και δεν φαντάζομαι ότι ε, θα σας εκπλήξει, γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ μικρή αλλαγή ένα ελάχιστο σφάλμα, ε, η λέξη corruption, την οποία εντοπίσαμε. Και έτσι θα υπάρξει μια διαφορετική διατύπωση. Ουσιαστικά το περιεχόμενο του φακέλου παραμένει άψεγάδιαστο θα έλεγα, άψογο και μπορούν τα κράτη-μέλη ε, του Συμβουλίου να το αποδεχθούν. Και χαιρόμαστε που έχουμε αυτού του είδους την πρόταση ενώπιον. Σας ευχαριστώ. Thank you very ευχαριστώ πολύ. Ιδίως ε, για το σχόλιο που είπατε ότι πόσο σας άρεσε αυτός ο κώδικας τη θεωρήσης. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μισελ να πω ότι μόλις ενημερωθήκαμε για το ότι δεν υπάρχει σήμερα δυνατότητα για διερμηνία από τα ρουμανικά και προς τα ρουμανικά. Δυστυχώς το πληροφορηθήκαμε πολύ λίγο πριν την συνάντηση και σας ζητώ συγγνώμη κύριε συνάδελφε, κύριε Άντζη. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ναι. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Λουί Μισελ, τον εισηγητή της Επιτροπής μας για το θέμα αυτό, για τον κανονισμό αυτό. Και εν συνεχεία, αν έχετε σχόλια ή συνάδελφοι, υπάρχει κάποιος χρόνος για συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άκρος ακριβή και λεπτομεριακή παρουσίαση αυτής της πρότασης τροποποίησης, γιατί περί αυτού πρόκειται όπως ακούσατε, μια περιορισμένη σε εύρος τροποποίηση του κώδικα θεωρήσεων. Διευκρινίστηκε αυτό. Πράγματι πρόκειται για μια τεχνική διόρθωση διατάξεων που αφορούν ε, τις θεωρήσεις για αεροδιαμετακόμιση. Και θα ήθελα να πω ότι με την ε, τροποποίηση αυτή δεν αλλάζει η πρακτική των κρατών μελών. Αυτό πρέπει να το υπενθυμίσουμε, είναι σημαντικό. Η τροποποίηση του κανονισμού λοιπόν προβλέπει ότι οι πήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι θεώρησης διαβατηρίου ή ε, έγκυρης άδεια παραμονής που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος το οποίο δεν εφαρμόζει ή δεν εφαρμόζει ακόμη εξ ολοκλήρου τις διατάξεις Σέγγεν Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, αυτές είναι οι χώρες, εξαιρούνται από την ε, υποχρέωση να έχουν στην κατοχή τους θεώρηση για την αεροδιαμετακόμιση. Έτσι ένα άτομο, Παραδείγματο χάρη Ιρακινής ποικότητα που έχει ε, έρχεται στην Βουλγαρία θα χρειάζεται, δεν θα χρειάζεται να έχει την δική αυτή θεώρηση ε, για αεροδιαμετακόμιση. Ένα άτομο το οποίο ήδη έχει θεώρηση ή άδεια διαμονής και το οποίο δηλαδή ήδη έχει ελεγχθεί εκ των προτέρων και επομένως έχει αναγνωριστεί ότι δεν ε, συνιστά κίνδυνο ε, λαθρομετανάστευσης θα μπορεί να απαλλάσσεται αυτή την υποχρέωση και έτσι απαλλάσσονται και από ένα επιπλέον διοικητικό άχθο και τα κράτη-μέλη, οι διοικήσεις των κρατών μελών. Εγώ προσωπικά, επειδή πρόκειται για τεχνική διόρθωση μεν, αλλά η οποία θα έχει και κάποια επίπτωση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ανθρώπους ουσιαστικά, έτσι, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Είμαι λοιπόν ε, υπέρ ε, της ε, γρήγορης, στο δυνατόν ταχύτερης διεκπαιρέωσης του θέματος Αφού δεν υπάρχει πρόβλημα, το είπε και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, νομίζω ότι καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε η πρόταση αυτή να έχει ευοδοθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Τώρα, θα μπορούσε να ψηφιστεί πριν τα τέλη του έτους. Από ό,τι μου λέει η γραμματεία, είναι λίγο ωριακό να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Πάντως, θα ήθελα να προχωρήσουμε το γρηγορότερο δυνατόν. Είπε και ο εκπρόσωπος τη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ουσιαστικά δεν έχει να κάνει με την αναθεώρηση του κώδικα θεωρήσεων που θα επανεξεταστεί μετά από 1,5 χρόνο ή 2 χρόνια. Άρα, αφού δεν συνδέονται αυτά τα δύο, γιατί να καθυστερήσει η διόρθωση αυτή. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο, γιατί νομίζω ότι πολύ συγκεκριμένα ε, υπόθηκαν όλα από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν προηγουμένως. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Δύο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ζόμερ και Άντζου. Ähm, Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οι ερωτήσει μου ουσιαστικά έχουν απαντηθεί από τα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε αυτό το λάθος και θα με ενδιέφερε και θα έπρεπε να είχε προσεχθεί αυτό. Και καλό είναι να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τι γίνεται με τις εκτελεστικές διατάξεις και το σχέδιο νόμου και τι γίνεται στην πρακτική εφαρμογή. Θα έπρεπε να είχε προσεχθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ουσιαστικά μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει προφανώς αυτό το λάθος, μια και πρόκειται για λάθος. Θα με ενδιαφέρε να άκουγα τα σχετικά πως έχουν και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου ολοκληρώνοντας είπε από πλευράς του ότι είναι ικανοποιημένος λέει το Συμβούλιο είναι ικανοποιημένο δύο φορές ασχολήθηκε με αυτό το θέμα όμως θα ήθελε κάποια άλλη διαφορετική διατύπωση αν κατάλαβα καλά ωραίο θα ήταν αν το Κοινοβούλιο ως το άλλο ίμιση του νομοθέτη, εκτός αν έκανα λάθος, γιατί ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου κουνάει το κεφάλι του τώρα. Μπορεί να επανορθωθεί αυτό. Ίσως δεν το κατάλαβα καλά με την άλλη διατύπωση. Τι εννοούσε. Όπως και οι προλαλήσαντες και οι προλαλήσασες, ε, πρόκειται για τεχνική υφή αλλαγές ή προσαρμογές. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Όμως έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από ό,τι κατάλαβα θα πρέπει παράλληλα με αυτές τις ε, τεχνικές τροποποιήσεις κάτι παραπάνω να διαγραφεί, δηλαδή η αναφορά σε σχέση με ημερομηνίες συνθήκων όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, τον ΕΟΧ. Γιατί να γίνει αυτό, θα ήθελα να μου δώσετε την απάντηση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ζητήσουμε στο τέλος να απαντήσει η Κομισιόν και Συμβούλιο. Κύριο Αντσούταρ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω γαλλικά. Αφού η Ρουμανία δεν έγινε δεκτή στο χώρο Σέγγιν δεν μπόρεσε να έρθει και μεταφραστής εδώ, διερμηνέας. Έμεινε στα σύνορα. Εντάξει, αστείο είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων. Τι θα ήθελα να πω. Λοιπόν, νομίζω ότι πέραν των τεχνικών τροποποιήσεων που προτείνονται, ουσιαστικά δίνεται και ένα συμβολικό μήνυμα. Δηλαδή, όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να την χάνουν ισότιμης μια διακριτικής μεταχείρισης. Είτε είναι μέλη του χώρου Σέγγεν, είτε δεν είναι. Νομίζω ότι είναι και ένα ε, δίδαγμα για τις διαδικασίες ένταξης ε, της Ρουμανία και της Βουλγαρίας ε, στην περιοχή Σέγγεν ή ευρύτερα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της διαχείρισης του χώρου Σέγγεν. Δεν θα πρέπει σε αυτήν την περίπτωση να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά λοιπόν. Νομίζω ότι οι τεχνικές τροποποιήσεις είναι φυσιολογικές και τις υποστηρίζουμε. Ώστε όλα να είναι σωστά και όπως πρέπει σε αυτόν τον κώδικα θεωρήσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω πραγματικά να μην υπάρχει συμβολικό ε, μήνυμα, να μην φτάνει τόσο μακριά αυτό το ε, γεγονός της έλλειψης ε, Ρουμάνων διερμιών σήμερα εδώ σε αυτή την αίθουσα. Ναι, θα ήθελα και εγώ να κάνω. εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις και όσον αφορά την παρουσίαση και από πλευρά του Συμβουλίου απαντήθηκαν ήδη νομίζω. Υποστηρίζουμε λοιπόν έτσι όλες τις προτάσεις και θα βοηθήσει ελπίζουμε αυτό τους ταξιδιώτες και θα τους διευκολύνει. Δρα, δρα, δρατώμενοι της ευκαιρίας θα ήθελα να σας αναφέρω το ίδιο το βίωμά μου την εμπειρία μου επιστρέφοντας πριν από μία εβδομάδα από το Στρασβούργο στη χώρα μου έπρεπε μια και υπήρχαν καιρικέ συνθήκε που παρακόλλιαν μέσω ενό αεροδρομίου που δεν είχε ζώνη τράνζιτ και έπρεπε να περάσουμε εκτός. Κάποια προβλήματα υπήρχαν και ίσως ελπίζω ότι η Κομισιόν θα το λάβει αυτό υπόψη. Ευχαριστώ. Thank you παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλά και μόνο να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για τις σαφέστατες επεξηγήσεις τους και να πω ότι ολόθυμα συμφωνώ με τις διεργασίες που εξηγήθηκαν από τον εισηγητή θα είχε ενταχθεί στο Σέγγεν η Κύπρος αν δεν υπήρχαν οι δυσκολίες που προκαλούνται από τον διχασμό την κατάσταση κατάληψη, την κατοχή της Κύπρου, του ημίσεως της Κύπρου. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό είναι μια τροποποίηση, μια αλλαγή που επανορθώνει τα πράγματα και την υποστηρίζουμε ως ομάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βλέπουμε ότι υπάρχει ευρύτατη υποστήριξη, αλλά υπήρχαν κάποια ερωτήματα και ζητήθηκε κάποια αποσαφήνιση από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή. Σας δίνω τον λόγο πρώτα στην Επιτροπή και μετά στο Συμβούλιο να αποσαφηνίσετε, να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Ποιος ε, είναι υπεύθυνο για το σφάλμα αυτό. Εγώ θα έλεγα να μην χάσουμε χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να πει ότι εμεί διατυπώσαμε την πρότασή μα, ε, ίσω οι συνομοθέτε, ε, οι γλωσσομαθεί νομικοί είναι υπεύθυνοι, που είναι απόντε, άρα δεν μπορούν να υπερασπίσουν αυτού εδώ. Λοιπόν, δεν είναι γνωστό ακριβώ το τι, προ... πρόβλημα προέκυψε, αλλά κάποια στιγμή όταν γίνεται το λεγόμενο χτένισμα του κειμένου, εκεί έγινε κάποιο λάθος, σε κάποιο σημείο θελήσαμε να υπάρχει υπάρχει μια συνοχή εκεί όμως που οι δύο έννοιες είχαν ε, διαφορετική σημασία. Δεν έχει όμως πλέον νόημα να αναζητήσουμε τον ένοχο. Τώρα, η αναφορά ε, στην Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ναι, τώρα μπορεί να διαγραφεί, γιατί στο άρθρο 3, όπως πλέον αναδιατυπώνεται με βάση την πρόταση, καλύπτονται πλέον όλα τα κράτη-μέλη, είτε είναι μέλη Σέγγεν ή μάλλον ε, είτε εκτός Σέγγεν, όπως είναι η Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, ή κράτη-μέλη που θα ενταχθούν στο Σέγγεν, αλλά όχι ακόμη, δεν είναι ακόμη σήμερα στο Σέγγεν. Και με την έννοια κράτος μέλος Σέγγεν καλύπτονται και οι συνδεδεμένες χώρες όπως η Ισλανδία. Επομένως δεν υπάρχει πλέον ανάγκη με τη διατύπωση που έχει αναθεωρηθεί όπως προτείνεται από την Κομισιόν δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να γίνεται αναφορά στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Ό,τι καλύπτεται από αυτή την έννοια πλέον ε, καλύπτεται με τη νέα διατύπωση. Άρα είναι περιττό πλεονάζει να αναφέρεται αυτή η συμφωνία. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ και πολύ σύντομα θα ξαναδώσω το λόγο στον πρόσωπο τη Πολωνική Προεδρία. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ζόμερ για το πολύ εύστοχο ερώτημά τη. Και μπορώ να σα πω ότι θα γίνει και ε, επισήμω. Θα σας πούμε, στο επίπεδο του Κορεπέρ θα εγκριθεί, αλλά το έχουμε ε, πει και στην Κομισιόν. Μόλις αντοπίσαμε μια τεχνική διόρθωση που πρέπει να γίνει στο προήμιο, στα σημεία 10 και 11 του κειμένου που γίνεται αναφορά στα άρθρα 3, 2 και 4, 2 ε, της Συμφωνίας ένταξη του 2005. 3-1-4-1 ε, θα έπρεπε να αναφέρεται στο κείμενο. Τεχνική παρατήρηση. Όταν είπα λοιπόν ότι διαφέρει διατύπωση, αυτό εννοούσα να αναφερόμαστε στα σωστά άρθρα της πράξης προσχώρησης. Περί αυτού μόνο πρόκειται. Επίσης το άρθρο 1 ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο είναι το σημαντικό που είναι και η ουσία της πρότασης και αυτό παραμένει ως έχει. Η πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επανέλθει ο εισηγητής μας ο κύριος Μισελ. Κοιτάξτε, πολύ σύντομα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο αλλά και τους συναδέλφους ε, για την υποστήριξή τους. Από ό,τι φαίνεται Υπάρχει πλήρης υποστήριξη από όλε τι πλευρέ σε αυτή την τεχνική διόρθωση. Θα υποβάλω λοιπόν ε, στα μέλη τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ πολύ σύντομα ένα σχέδιο έκθεση που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε πολύ γρήγορα στο πλαίσιο μια ε, συνεδρίασής μα. Εγώ θα έλεγα αν είναι δυνατό στα τέλη Νοεμβρίου, ούτω ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τάχιστα. Και αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε, αφού φαίνεται ότι υπάρχει συνένεση, ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε και να διορθώσουμε αυτό το τεχνικό σφάλμα. Να το αφαιρέσουμε από την νομοθεσία μα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία μέχρι τα τέλη του έτους όπως ζητεί και ο εισηγητής μας. Μπορούμε λοιπόν τώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο, το οποίο αφορά την τροποποίηση του κανονισμού όσον αφορά τη συμπερίληψη της περιοχής του Καλίνικρατ και ορισμένων πολωνικών νομών στην επιλέξιμη παραμεθόρια περιοχή. Η συγκεκριτής μας είναι ο κύριος Τρενταφυλλίδης. Θα σας δώσω το λόγο κύριε Ισηγητά και εν συνεχεία θα μιλήσουν οι πρόσωποι Κομισιόν και Συμβουλή και θα ακολουθήσει συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όπως και το προηγούμενο θέμα, αυτή η έκθεση είναι απλή υπόθεση και χωρίς προβλήματα. Στόχος μας είναι να αρθούν τα προσκόμματα και εμπόδια σε πολύχρονους δεσμούς όσον αφορά τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Καλίνιγκρατ και Μαζούρσκι που με την ε, διεύρυνση του 2004 και με την τροποποίηση του κανονισμού όσον αφορά τις μεθοριακές αυτές ε, επαφές ε, και όσον αφορά τα σύνορα καθορίζοντας τοπικών σύνορων περιοχές. Η τροποποίηση προβλέπει μια εξαίρεση στον κανονισμό επιτρέποντας το σύνολο του όμπλαστ της περιφέρειας Καλίνιγκραντ και της ευρύτερης περιοχής με τα σύνορα με την Πολωνία να θεωρείται μεθοριακή περιοχή ώστε να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό υφιστάμενων περιοχών και να διασφαλίσουμε ότι οι κάτοικοι αυτή τη ευρύτερη περιοχή θα μπορούν να μετακινούνται εύκολα χωρί να προσαρμόζονται σε διαφορετικέ απαιτήσει. Υποβάλλεται αυτή η πρόταση λόγω των διαφορετικών πρωτοβουλειών που έχουν αναλυθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων του Καλίνιγκραντ, όπως ε, το μέσο του, της θεώρησης διαβατηρίου και το 2000, του 2007 η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας που δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την περιθωριοποίηση του Καλίνιγκρατ και των κατοίκων του. Είμαστε ε, ικανοποιημένοι για αυτήν την τροπολογία για διάφορους λόγους. Πρώτον, διευκολύνει την κίνηση, τη μετακίνηση πολιτών από την ίδια περιοχή προς τα Πέριξ. Ενισχύει τις γειτονικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών στα εξωτερικά σύνορα και συνεισφέρει φυσικά σε ένα χώρο ελευθερίας και ευημερίας πέρα από τα ίδια τα σύνορα της ΕΕ. Και αυτό είναι ο λόγος, ε, συνάδελφοι, για τον οποίο αποφάσισα να μην καταθέσω τροπολογίες. Ευχαριστώ. And Σας ευχαριστώ. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει τον λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ. Ευχαριστώ, θα είμαι συντομοτάτη. Η πρόταση αυτή είναι πολύ θετική, είναι συμβατή με την πρόταση της Επιτροπής. Επιβεβαιώνουμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτή είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση η οποία δεν δημιουργεί κανένα προηγούμενο για αδίποτε τέτοια πρόταση στο μέλλον. Ευχαριστώ για το σχόλιο σας. Το λόγο στην Πολωνική Προεδρία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έρχομαι εδώ σήμερα για δεύτερη φορά, παίρνω το λόγο, και θα με ακούσετε κι άλλο γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία ε, θα κληθώ να σχολιάσω. Για το Καλίνιγκραντ τώρα θα ήθελα να σας ενημερώσω για το που βρισκόμαστε στις 27 Οκτωβρίου. Το Συμβούλιο συζήτησε το θέμα του Καλίνιγκραντ και γι' αυτό εδώ επιτρέψτε μου να μιλήσω σαν εκπρόσωπος της Προεδρίας αλλά να εκφράσω επίσης και την χαρά της πολωνικής πλευράς γιατί όλοι οι εκπρόσωποι και οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών κατανόησαν το θέμα και οι αρμόδιοι υπουργοί είπαν ότι θα πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα των bona fide καλή την πίστη ταξιδιωτών που μπορεί να χρησιμοποιούν τις τοπικές διευκολύνσεις ε, για τις μετακινήσεις τους στο μέλλον. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στους δύο φακέλους, τα δύο θέματα που είναι κρίσιμα για να κατανοήσει κανείς τις συζητήσεις στο Συμβούλιο τους τελευταίους δύο μήνες. Η πρώτη ρύθμιση είναι η κοινή δήλωση η οποία συμπεφωνήθη την προηγούμενη εβδομάδα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Σε αυτήν την κοινή δήλωση λέγεται ξεκάθαρα ότι τώρα πλέον έχουμε μπροστά μας μία εξαίρεση, μία εξαίρεση που δεν δημιουργεί προηγούμενο. Παρόλα αυτά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί, θα πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό εποπτείας ισχυρότατο και αυτό είναι τμήμα της λύσης που συμφωνήθηκε ανάμεσα στην Επιτροπή για τις χώρες μέλη. Το δεύτερο τμήμα είναι ότι η κοινή δήλωση η οποία παρουσιάστηκε από την πολωνική αντιπροσωπεία λέγει ότι θα πρέπει να ξεπεραστούν τα, τα, οι κανονικές, οι τακτικές ρυθμίσεις που προέρχονται από τον κανονισμό και εδράζονται στον κανονισμό του 2006. Γι' αυτό η διεύρυνση αυτή δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι είναι εμπόδιο σε αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με την προστασία των πολιτών. Η λύση αυτή πάντως παραμένει μία εξαίρεση. Όπως το είχα πει και την προηγούμενη φορά είμαι στην διάθεσή σας και αν έχετε κάποιες ερωτήσεις με τις οποίες μπορώ να βοηθήσω είμαι ξανά στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν το κατάλαβα ότι μου δώσε τον λόγο. Είμαι σκιώδη εισηγητής. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τον κύριο Κυριάκο Τριανταφυλλίδη, επειδή έκανε πολύ καλή δουλειά. Παρότι το θέμα φαίνεται περιορισμένης εμβέλειας. Παρόλα αυτά, η προσθήκη της περιοχής του Καλίνγκαρτ και κάποιων περιοχών της Πολωνίας ω μεθοριακών, όχι μόνο θα είναι καλό για του πολίτε του Καλίνιγκρατ, αλλά είναι επίση πολύ σημαντικό για την οικονομία τη ευρύτερη περιοχή και αυτό είναι πρόδειλο, είναι προφανέ. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε απέναντί μα μια πραγματική πολιτική προσέγγιση ως πρωτοβουλία και πρέπει να υποστηριχτεί αυτό. Είναι πολύ καλό λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών προκατακτικών εργασιών είχαμε καλή συνεργασία και σαν αποτέλεσμα αυτού έχουμε την υποστήριξη πλήρως της έκθεσης. Δεν έχουμε πρόθεση να καταθέσουμε καμιά τροπολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μπουσετήλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Απλώς και εγώ να πω ότι από πλευρά του ΕΡΚ υποστηρίζουμε αυτή την έκθεση και το έργο του κυρίου Τριανταφυλλίδη και εμείς. Και εμείς επίση συμφωνούμε ότι αυτό το ένα εκατομμύριο κατοίκων στο Καρλίνιγκρατ πρέπει να αποφύγει την απομόνωση, την περιθωριοποίηση και γι' αυτό δεχόμαστε αυτή την πρόταση. Ακόμα και ικανοποιεί και την πολωνική αντιπροσωπεία. Γιατί να μην το υποστηρίξουμε λοιπόν. Ευχαριστώ. πρόεδρο, ευχαριστώ. Κυρία Ζανόκα, παρακαλώ. Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται η συζήτηση αυτή. Εμείς υποστηρίζουμε πλήρως uh, τη συγκεκριμένη πρόταση Είμαστε μέλος της αντιπροσωπείας με την Ρωσία, επισκεφθήκαμε την περιοχή, είδαμε τα προβλήματα στα σύνορα, γι' αυτό με ρεαλιστικό τρόπο διευκολύνεται η κατάσταση. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα σχόλια μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν δημιουργείται κάποιο άλλο θέμα. Το επόμενο θέμα μας λοιπόν για μια στιγμή. Μια στιγμή. Η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Τετάρτη 9η Νοεμβρίου. Και εδώ μου λένε ότι οι τροπολογίες θα πρέπει να, σταλούν στην γραμματεία με μορφή Word και όχι με οποιαδήποτε άλλη μορφή. Ελπίζουμε να φτάσουμε έτσι στην Ολομέλεια τον μήνα Δεκέμβριο. Περνάμε στο σημείο 5 τώρα για την κατάργηση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγητής μας, η συγγήτριά μας είναι η κυρία Στάνουκα και θα της δώσω το λόγο για να παρουσιάσει την έκθεσή της κυρία Στάνουκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας στις εκθέσεις της Επιτροπής Αναφορών. Είμαι μέλος άλλωστε και της Επιτροπής Αναφορών. και είμαι σκιώδης εισηγήτρια για την έκθεση της κυρίας Βαλεάν για την πολιτική μου ομάδα. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια και για την Επιτροπή μας. Ελπίζω η συνεργασία μας να είναι καλή. και να <clears throat> παρουσιαστούν κάποιες αρκετά χρήσιμες προτάσεις. Έξι σημεία περιλαμβάνει η γνωμοδότηση. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει σταθεί ιδιαίτερα δραστήρια στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτό. Δεν έχει αντιμετωπίσει ε, τις παραβιάσεις, σαν παράδειγμα, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λειτουργήσει περισσότερο προληπτικά. Υπάρχει το πρόβλημα της ελεύθερης διακίνησης, είναι σαφές. Αυτό το βλέπουμε στο σημείο 3 περισσότερο. Εκφράζουμε άλλωστε και την ανησυχία μας για την ελληματική εφαρμογή της οδηγίας, που είναι οδηγία όπως έχουμε πει για την ελεύθερη διακίνηση. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα δυστυχώς στην ελεύθερη διακίνηση και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών και γι' αυτό καλούμε όλες τις πλευρές να μεταφέρουν σωστά το κοινοτικό κεκτημένο στην ομοθεσία τους. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η άσκηση του δικαιώματος ψήφου. Συμμετοχή στην ψηφοφορία. Ξέρετε ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μένουν σε μια άλλη χώρα έχουν θεωρητικά το δικαίωμα συμμετοχή στις ευρωπαϊκές και στις τοπικές εκλογές. Υπάρχουν όμως παρόλα αυτά αρκετά προβλήματα. Η εφαρμογή συνεπώς των συγκεκριμένων δικαιωμάτων πρέπει να επανεξεταστούν γιατί είναι πολύ λίγοι οι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι ασκούν το δικαίωμα ψηφοφορίας στην χώρα παραμονής τους. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υπάρχουν προβλήματα και τεχνικά και γραφειοκρατικά. Γι' αυτό ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να διευκολύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στις τοπικές και ευρωπαϊκές εκλογές. Ένα άλλο θέμα είναι τα δικαιώματα των ανθρώπων των απάτριδων που δεν έχουν εν πάση περιπτώσει την ιδιότητα του πολίτη ενός κράτους και σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν να παίρνουν μέρος σε κάποιες από τις εκλογικές διαδικασίες. Ζητούμε λοιπόν από τα ευρωπαϊκά όργανα και τα κράτη-μέλη να ορίσουν σωστά τα δικαιώματα των πολιτών που προέρχονται από τρίτες χώρες με τα δικαιώματα των πολιτών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητάμε επίσης από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις των εθνικών οργανισμών που ασχολούνται με την ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων αυτών ιδιαίτερα του δικαιώματος της συμμετοχής στις τοπικές εκλογές, του εκλέγειν, μάλλον στις τοπικές εκλογές. Στο σημείο 5 έχουμε την άσκηση του δικαιώματος προξενικής προστασίας όταν έχουν ανάγκη από μια τέτοια μορφή προστασίας οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχει το αντίστοιχο προξενείο σε μια άλλη χώρα, τότε σε αυτή την περίπτωση διατηρούν το δικαίωμα της προξενικής προστασίας από ένα άλλο κράτος μέλος το οποίο έχει αυτές τις εγκαταστάσεις. Λοιπόν, αυτές είναι οι βασικές προτάσεις που περιλαμβάνει η έκθεση. Προτείνουμε να υπάρξει μια γνωμοδότηση λοιπόν, η οποία να εφαρμόσει, να περιλαμβάνει τις προτάσεις μάλλον της Επιτροπής Αναφορών. Καλώς λοιπόν σχόλια, ερωτήσεις, η κυρία Σώμα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα όμως κάποια σχόλια να κάνω στην έκθεση αυτή. Και πρόκειται για το εξής. Πιστεύω ότι το θέμα είναι η έκθεση για την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπάρχουν λιγότερα εμπόδια για τα δικαιώματα της ηθαγένειας, για τους πολίτες όμως της Ένωσης, αν το κατάλαβα καλά. Τότε θα έλεγα ότι κάποια πράγματα δεν έχουν θέση, δεν έχουν θέση σε αυτή την έκθεση. Το σημείο 2 όπου πρόκειται για τους απάτριδες για παράδειγμα. Δεν έχει θέση εδώ. Δεν έχει καμιά σχέση με τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέμα των απάτριδων. Και για την τελευταία περίοδο στο 1 για υπηκόους τρίτων χωρών με μόνιμη έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσαρμοστούν στα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα δικαιώματά τους. Ακούστε, πολύ επικίνδυνο αυτό. Εγώ θα έλεγα δεν μπορούμε να το δεχτούμε κάτι τέτοιο ως αίτημα. Τώρα, από την άλλη μεριά, το 3, το σημείο 3 <coughs> για την ε, ανεπαρκή εφαρμογή της οδηγίας ιδιαίτερα όσον αφορά την οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία Μάλιστα. Και κυρίως για την οδηγία περί υπηρεσιών. Όμως δεν έχει και μεγάλη σχέση με τη δική μας επιτροπή αυτό το θέμα. Παρόλα αυτά. Στο σημείο 4 τώρα. Στο σημείο 4 εκπροσωπεί την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να ώστε οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν σε ένα άλλο κράτος μέλος εκτός του δικού τους να μπορούν να συμμετέχουν στις περιφερειακές εκλογές, ευρωπαϊκές εκλογές, δημοτικές εκλογές. Δεν ξέρω τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι έργο των κρατών μελών αυτό και όχι της Επιτροπής, των περιφερειών αλλά των δήμων και κοινοτήτων κυρίως που διοργανώνουν τέτοιες ε, εκλογές. Να αλλάξει ίσως λοιπόν αυτό το εδάφιο, να τροποποιηθεί. Και στο σημείο 6 ομολογώ ειλικρινά είναι πολύ γενικόλογο και αφηρημένο αυτό και θα έλεγα ότι είτε πιο συγκεκριμένα χειροπιαστά παραδείγματα πρέπει να αναφέρουμε ή τέτοια συλλήβδην κρίση θα πρέπει να την αποφύγουμε, να την αφήσουμε εκτός μια τέτοια συνολική κρίση. Ευχαριστώ. Thank you Σε ευχαριστούμε. Και κάποια άλλα σχόλια από τον κύριο Ιτσεφ πρώτα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ω σκιώδης εισηγητής για την ομάδα Άντε θα παρέμβω και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία εισηγήτρια για το έργο της. Μεταξύ των πολλών σημαντικών σημείων θα ήθελα να αναφερθώ στο σημείο 3. Πρώτα απ' όλα, περίπου 25% του συνολικού αριθμού των αναφορών που υποβάλλονται αφορούν προβλήματα ελεύθερης κυκλοφορίας. Προφανώς διαρκώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα τους επόμενους μήνες και έτη. Όλο και περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες και επειδή δεν τηρούνται οι οδηγίες και κανονισμοί οι, οποίες έχουν ήδη, και οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί. Θέλουμε να ζητήσουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυ σε αυτήν την υπόθεση και στην έκθεση, στην ολοκλήρωση της έκθεσης θα είναι μια πολύ καλή αφορμή για να ενταθούν οι προσπάθειες με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάποια κράτη-μέλη φέρονται σαν να μην υπάρχει καν οδηγία περί ελεύθερης κυκλοφορίας πολιτών. Δεν σέβονται αυτή την ε, ε, οδηγία. Γι' αυτό πρέπει τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα να ενεργοποιηθούν δραστήρια για τα δικαιώματα των πολιτών και της κοινωνίας. Δυστυχώς βλέπουμε μια φθήνουσα τάση όσον αφορά τα κράτη-μέλη σε σχέση με το σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών. Και σε αυτή την πτυχή αποστέλει ένα έντονο μήνυμα προειδοποίηση, συναγερμού η έκθεση για τους Ρωμά, για τους Τσιγκάνους δεύτερο. Πάλι αυτό το θέμα εκκρεμεί στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές προσπάθειες πρέπει να γίνουν για τη στέγαση, εκπαίδευση, κατάρτιση, ελεύθερη κυκλοφορία των συγκάνων. Και τα κράτη-μέλη πρέπει να μεριμνήσουν για την κοινωνική ένταξη και στην κοινωνία και τις κοινωνίες των παιδιών των συγκάνων. Οι προειδοποιήσεις από την έκθεση αναφέρουν ότι το θέμα των Ρωμά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με θετικό τρόπο υπό προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζονται τα δικαιώματα των συγκάνων με ίση βάση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης η πληροφόρηση για τα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες. Ένας μεγάλος αριθμός πολιτών που ζουν σε κράτος εκτός του δικού τους δεν έχουν πλήρη πληροφόρηση για το ποια δικαιώματα έχουν. Πρέπει να διευρύνουν αυτό το σύστημα πληροφόρησης για αυτούς τους ανθρώπους τα κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα όσον αφορά εκεί που αντιμετωπίζουν προβλήματα και όσον αφορά περιορισμούς δικαιωμάτων, κοινωνικά δικαιώματα, υγεία, υγειονομικά θέματα καταναλωτών, δικαιώματα κτλ. Ακόμα παραπάνω, οι υφιστάμενες διοικητικές διατάξεις και διεργασίες σε πολλά κράτη-μέλη είναι τόσο χρονοβόρες που καμιά φορά είναι εξισούνται, εξισώνονται με άρνηση δικαιωμάτων για αυτούς τους πολίτες. Πρέπει αυτή η γραφειοκρατική επιβάρυνση λοιπόν να αντιμετωπιστεί και αυτοί οι περιορισμοί να αντιμετωπιστούν. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα που θα καταθέσω τροπολογίες και ελπίζω ότι με τη βοήθεια όλων των συναδέλφων θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κατάσταση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων λαμβάνοντας πολύ υπόψη αυτά τα θέματα της έκθεσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Φάνο, επόμενα μιλήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία έχουν πει οι προλαλήσαντες, ιδιαίτερα ο συνάδελφος Λίτσεφ. Ευχαριστώ την κυρία Ζανόκα για την πρότασή της βέβαια. Θα ήθελα όμως να πω ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε το σημείο 3 για την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οικογενειών τους. Όπως είπε ο συνάδελφος Σίλτσεφ, υπάρχουν κάποια προβλήματα με τους Ρώμ στο συγκεκριμένο, με τους Ρωμά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και όχι μόνο, αλλά και ε, με τους ε, E io in questo ritengo che Υπάρχουν προβλήματα και στην ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων πολιτών με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα καταθέσω ορισμένες τροπολογίες προς την κατεύθυνση της κάλυψης των αναγκών των πολιτών με διαφορετικό ε, σεξουαλικό ή γενετήσιο προσανατολισμό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, διάβασα προσεκτικά τη γνωμοδότηση και θα ευχαριστήσω την συγγραφέα για αυτόν τη γνώμη που έχει εκφράσει. Και εγώ όταν διάβαζα είχα επικεντρωθεί πιο πολύ στα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και όχι των πολιτών τρίτων χωρών. Γιατί υπάρχουν πολλές άλλες οδηγίες για τους πολίτες τρίτων χωρών αντιλαμβάνομαι ότι η συγκεκριμένη οδηγία θα πρέπει να επικεντρωθεί πιο πολύ στο δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να διακινούν ελεύθερα και εκείνο το οποίο εντοπίζει η έκθεση 2010 για την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι οι ίδιοι Ευρωπαίοι πολίτες όταν ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από το κεκτημένο της ενιαίας αγοράς πολλές φορές αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια είτε είναι οικονομικοί φορείς, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι καταναλωτές, είτε είναι εργαζόμενοι. Και ο, ο είναι ακριβώς να βρεθούν ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και να τα υπερπηδήσουμε. Ε, επίσης υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά... Ε, δεν είναι πρόβλημα η έλλειψη νομοθεσίας. Το πρόβλημα είναι η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας που υπάρχει Πώ διασφαλίζει στου ευρωπαίου πολίτε να απολαμβάνουν τα δικαιώματά του. Και εκείνο το οποίο προκύπτει από την έκθεση του 2010 είναι ότι οι φυστάμενοι κανόνε είτε πρέπει να επεκταθούν και να επικαιροποιηθούν, είτε να επανεξεταστούν ριζικά ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε τις διάφορες κοινωνικο-οικονομικές ή τεχνολογικές πραγματικότητες και να προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των Ευρωπαίων. Ε, οι πολίτες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα. Ε, εγώ είμαι συγκήτρια για την έκθεση που αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος 2013 για τα δικαιώματα των πολιτών και πιστεύω ότι πρέπει να δούμε περισσότερο πώς ο Ευρωπαίος πολίτης να γνωρίζει τι του προσφέρει η ηθαγένειά του και να αποκτά τα δικαιώματα στην πράξη, όχι απλά να έχει άγνοια για τα συγκεκριμένα και επίσης πώς να πλουστεύσουμε στην άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων κάθε πολίτη στην καθημερινότητά του, γιατί εκείνη που αντιμετωπίζει προβλήματα. Πρέπει να πω ότι όταν μιλούμε για τα δικαιώματα των τρίτων χωρών, τα σέβομαι απόλυτα, αλλά ας επικεντρωθούμε και λίγο στα δικαιώματα Ευρωπαίων πολιτών που στερούνται το δικαίωμα να διακινούνται ελεύθερα. Μιλώντας για τη δική μου τη χώρα, την Κύπρο, το δικό μα δικαίωμα να διακινούμαστε ελεύθερα που είναι αναφέρει το δικαίωμα κάθε Ευρωπαίου πολίτη, το στερούμαστε. 37 ολόκληρα χρόνια δεν μπορούμε να διακινηθούμε ελεύθερα στο νησί. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να το φέρω ενώπιον τη, στη γνώση των συναδέλφων. Διότι δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι στην Κύπρο δεν μπορεί εγώ, ο Ευρωπαίο πολίτη, να διακινηθώ ελεύθερα από άκρη σ' άκρη στο νησί. Έχω περιορισμού. Επομένω, κάθε φορά που γράφω γνωμοδοτήσει ή ασχολούμαι με τα δικαιώματα των ατόμων από τρίτε χώρε, ειλικρινά νιώθω ότι υπάρχει μια τραγική ηρωνία. Γιατί και δικαιώματα Ευρωπαίων πολιτών καταπατούνται και εδώ πρέπει να το έχουμε υπόψη μα. Εγώ προσωπικά θα κάνω κάποιε τροπολογίε, δίνοντα έφαση κυρίω στην καλύτερη ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών, ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά του και στην πράξη να τα διεκδικούν και να εφαρμόζονται. Ευχαριστώ. Thank you very much. And... Σας ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ήθελα απλώς να ευχαριστήσω την κυρία Ζτανόκα για την έκθεσή της. Ε, να πω ότι μαζί με την συνάδελφο που είναι σκιώδης ε, εισηγήτρια από την ομάδα μου θα δούμε με λεπτομέρεια κατά πόσο θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες αλλά εκ πρώτης όψεως θέλω να πω ότι οι εισηγήσει που γίνονται σε αυτό το κείμενο τις βρίσκω να είναι προς την ε, ορθή κατεύθυνση και μάλλον η ομάδα μου θα στηρίξει την έκθεση όπως θα διαμορφωθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους ε, για τα σχόλιά σας. Έχετε και κάποιες προτάσεις ε, που θα πρέπει να διανεμηθούν για να δούμε αν θα μπορέσουν να συμπεριληφθούν ή όχι. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Στανόκα, η οποία θα δώσει τις απαντήσεις της. Yes. Ε, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χειώδες εισηγητές, αλλά και όλους τους άλλους συναδέλφους για τις προτάσεις τους. Σας ευχαριστώ λοιπόν και θέλω να σας πω ότι είμαι διατεθειμένη να συζητήσουμε και να συμπεριλάβω και τις τροπολογίες σας στο σύντομο αυτό έγγραφο. Πρώτα απ' όλα, ναι, πράγματι πρέπει I think... Ε, να δούμε και το θέμα των εποχιακών εργαζομένων στην ομοδότηση αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ελεύθερη ε, κυκλοφορία και το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης, προτάσεις σας ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες. Είναι μια γνωμοδότηση Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Για να αφορά σε άλλα δικαιώματα, όπως αυτά που ε, διέπονται από νοδία για τις υπηρεσίες ή άλλες οδηγίες, ελπίζω και αυτά όλα να συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο της έκθεσης, αλλά δεν είναι δικής μας ε, αρμοδιότητας ακριβώς. Δεν μπορούμε εμείς ως Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να κάνουμε αυτές τις συγκεκριμένε προτάσεις. Κάτι άλλο. Συμφωνώ και καλωσορίζω τις προτάσεις για την αναφορά συγκεκριμένα στο πρόβλημα των Ρωμά πράγματι πρέπει να αναφέρεται. καθώς και τα άτομα με διαφορετικό γενετήσιο ή σεξουαλικό προσανατολισμό. Αυτές οι δύο κατηγορίες πράγματι αντιμετωπίζουν ε, περισσότερα και συγκεκριμένα προβλήματα, ιδίως ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία ζευγαριών. Θα μπορούσαμε λοιπόν να το αναφέρουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το να φέρουμε υπηκόους ε, τρίτων χωρών, non-citizens ή third country citizens, εκεί που μιλάμε για third country nationals, για υπηκόους τρίτων χωρών, στον ορισμό εντάσσονται και οι αλλοδαποί αλλά και άτομα ε, που είναι απάτριδα, που δεν έχουν δηλαδή κάποια επικότητα. Υπάρχουν, ε, βέβαια σε αυτήν την περίπτωση μιλάμε μόνο για μονίμως διαμένοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατηγορίες αυτές λοιπόν φυσικά τα δικαιώματά τους καλύπτονται από την Οδηγία 189. Αλλά αν λέμε το δικαίωμα να είναι μονίμως διαμένοντες, να ενταχθούν στην κοινότητα, στην περιοχή, εδώ μιλάμε ουσιαστικά για τη συμμετοχή σε τοπικές εκλογές. Direction in which by my opinion κατά την ε, άποψη και τη δική μου και της ε, πολιτικής μου ομάδας ε, μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, μπορούμε να εξετάσουμε κάποιες προτάσεις, αλλά το σημείο αυτό ουσιαστικά αναφέρεται σε μια διαφορετική ιδιότητα υπηκόου, μια συγκεκριμένη κατηγορία υπηκόου. Μιλάμε για τα δικαιώματα για την Ευρωπαϊκή Θαγένεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναφέρονται και άλλοι μονίμως διαμένοντες ως υπήκοοι και θα πρέπει να υπάρχει η εναρμόση των δικαιωμάτων τους με τα δικαιώματα των υπηκών αυτών. Σε ό,τι αφορά τώρα την Κομισιόν, βεβαίως μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. στην Επιτροπή Αναφορών να την αντιμετωπίζουμε και εξετάζουμε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Όταν πολίτες ενός άλλου κράτους μέλους δεν μπορούν να ασχίσουν ελεύθερα το δικαίωμα του εκλέγην αν δεν ζουν στο κράτος ε, την υπηκότητα το οποίο έχουν, υπάρχουν προβλήματα πραγματικά και η Επιτροπή που είναι θεματοφύλακα των συνθήκων και στην προκειμένη περίπτωση αυτών των αυτών των δικαιωμάτων των πολιτών πράγματι πρέπει να φροντίσει μαζί με τα κράτη-μέλη να αντιμετωπιστεί τέλος πάντων να γίνει γνωστό αυτό το θέμα. Φυσικά και μπορούμε να το συζητήσουμε ε, την περαιτέρω αυτό το θέμα. Όπως σας είπα λοιπόν είμαι ανοιχτή, μπορώ να συζητήσουμε όλες τις τροπολογίες σας και θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Πράγματι, θα συζητήσουμε τα σχετικά θέματα. Έχει συζητηθεί και έχει ζήτηθει μάλλον από την Κομισιόν να αλλά βλέπω τη Σάρα Λάτφορντ να έχει σηκώσει το χέρι. Θέλετε να πείτε κάτι, κυρία Λάτφορντ, έχετε το λόγο. Λυπάμαι που έχασα την παρουσία της κυρίας Σανόκα. Κοιτάξτε, εμείς ήταν το τελικό της σχόλιο, εμείς κλείνουμε το θέμα. Είχα ζητήσει από την κυρία Σδενόκα να κλείσει τη συζήτηση. Α, ήρθα ακόμα πιο αργά από όσο νόμιζα. Ένα μικρό σχόλιο, επιτρέπετε παρακαλώ. Λοιπόν, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ζανέκα και την κυρία Βαλέαν στην Επιτροπή Αναφορών. Έχοντας δει την προσπάθεια που έχει γίνει στην Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις κάρτες παραμονής, σχετικά με τη χορήγηση των θεωρήσεων. Έρχομαι από το Ηνωμένο Βασίλειο και από το Λονδίνο συγκεκριμένα και υπάρχουν πολλές οικογένειες που ε, για να τους επισκεφθούν έχουν ανάγκη από βίζες τύπου Σέγγεν. Και έχω και πάρα πολλούς εκλογείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στα πλαίσια της αναγνώρισης των ε, κοινωνικών συμφωνιών συγκατοίκητης ή συμβίωσης ή και των γάμων μερικές φορές μεταξύ δύο ατόμων του ιδίου φύλου. Όλοι γνωρίζουμε το μέγεθος των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες μας. Και είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο να συμβαίνει το 2011. Τόσα χρόνια μετά από τον όρο της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη ή την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, αν θέλετε, ήδη από το 2006 υπάρχει πλήρης ε, ε, ελεύθερη διακίνηση, αλλά παρόλα αυτά τα εμπόδια είναι σημαντικά. Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη και γι' αυτό καλό θα ήταν να μπορέσουμε να αποδείξουμε στους εκλογείς μας ότι αυτό το τμήμα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος δουλεύει καλά, όπως είχε προβλεφθεί. Να ζητήσω λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γνωρίζοντας ότι προσπαθούν να περάσουν σε σωστή εφαρμογή, των κανόνων και ταυτόχρονα να ασκούν αυστήρα ε, τις διαδικασίες επί παραλήψη ή επί παραβάση σε σχέση με την εφαρμογή των κανόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται να φέρει εις θετικά την αποστολή της και να αναλάβει νομική δράση για να ξεπεραστούν τα εμπόδια, οι τροχοπέδες στην ελεύθερη διακίνηση ανεξαρτήτως ε, του καθεστώτος το οποίο χαρακτηρίζει ε, τους πολίτες οι οποίοι προχωρούν σε γάμους ιδίου φίλου σαν παράδειγμα και να μην λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ότι είναι θέμα εθνικών ευθυνών και εθνικών νομικών ρυθμίσεων. Όχι. Αυτό είναι δικαιολογία. Όλο ωραία λόγια ακούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καιρό είναι πλέον να ακούσουμε και πράξεις σε σχέση με την εφαρμογή των συγκεκριμένων κανόνων. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όλοι αναφερθήκατε στις ε, δυσκολίες που υπάρχουν για την εφαρμογή της οδηγίας για την ελεύθερη διακίνηση. Θα ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να μην μας πείτε μόνο λόγια, αλλά να μας δώσετε και στοιχεία για τις ενέργειες οι οποίες θα ακολουθήσουν. Κυρία Γεωργιάδου, αν άκουσα καλά. Ναι, πράγματι, όλη αυτή η ουσία της έκθεσης για την ηθαγένεια για τους πολίτες ήταν να ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και την άρση των προσκομμάτων που παρεμποδίζουν τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων τους. Σχεδόν 20 χρόνια πέρασαν και το 2015 θα είναι 20 χρόνια από την εισαγωγή αυτής της προσέγγισης των δικαιωμάτων της ηθαγένειας. Και αυτή η έκθεση ήθελε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώματά τους οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλωσορίζουμε λοιπόν και προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το εγχείρημα για να προαχθεί αυτή η πρωτοβουλία. Για τα συγκεκριμένα θέματα στο σχέδιο γνωμοδότησης. Πρώτα απ' όλα, έχει συνειδητοποιήσει σαφώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η κατάσταση ατόμων που ανήκουν σε μιονοτικές ομάδες και που ζουν σε κράτη-μέλη αλλά δεν έχουν την ηθαγένεια, την υπηκότητα αυτών των κρατών μελών είναι ένα πολύ ευαίσθητο, ακαθόδε θέμα. Φυσικά πρέπει να δοθεί ιδέουσα προσοχή στο γεγονός ότι οι όροι και προϋποθέσεις στο να πάρει κανείς την υπηκότητα ή να χάσει την υπηκότητα ενός κράτους μέλους ρυθμίζονται αποκλειστικά όλα αυτά τα θέματα από την ομοθεσία των κρατών μελών. Κάθε κράτο μέλο έχει την ελευθερία, διακριτική ελευθερία, να καθορίζει πώ απονέμεται η υπηκότητα ακόμα και σε απάτριδε και τι γίνεται σε σχέση με αυτού. Δεν έχει δικαιώματα να παρεμβαίνει σε αυτά τα θέματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τα κράτη-μέλη έχουν αποκλειστικά δικαιώματα να θεσπίζουν ρυθμίσεις και συμμετοχή για τέτοια άτομα που δεν έχουν την υπηκότητά τους και τη συμμετοχή τους σε δημοτικές και τοπικές εκλογές. Και πάλι, το ευρωπαϊκό δίκαιο ρυθμίζει τα θέματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν σε κράτος εκτός του δικού τους για να συμμετέχουν και να είναι και υποψήφοι σε τοπικές εκλογές και σε ευρωπαϊκές εκλογές ακόμα και αν δεν έχουν την υπηκότητα του κράτους στο οποίο κατοικοεδρεύουν. Θέματα όμως όσον αφορά τη συμμετοχή σε δημοτικές και τοπικές εκλογές για άτομα που δεν είναι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται εκτός ακριβώς του φάσματος του ευρωπαϊκού δικαίου. Και όσον αφορά τώρα την ε, συμμόρφωση, όσον αφορά και την επιβολή των δικαιωμάτων, αυτά απορρέουν από συνθήκη και από την Οδηγία για την Ελεύθερη Κυκλοφορία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί μια πολιτική αυστηρής εφαρμογής αυτών των διατάξεων. Μέχρι σήμερα είχαμε χειροπιαστά σημαντικά αποτελέσματα. Έχουμε διαθρωμένο, δομημένο διάλογο με τα κράτη-μέλη και τις περισσότερες φορές τροποποιείται ή βελτιώνεται η νομοθεσία ώστε να συμμορφώνεται άμεσα με την οδηγία περί ελεύθερης κυκλοφορίας και παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ αυτά τα τεκτενόμενα, ώστε τα κράτη-μέλη να έρθουν στο ύψο των δεσμεύσεών του και να συμμορφωθούν. Για όσα κράτη-μέλη δεν έχουν φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο, έχουμε ασκήσει προσφυγή περί παραβίαση ή παράβαση. Μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου είχαμε προσφύγει έναντι 12 κρατών μελών αφορούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, ακόμα και θέματα όσον αφορά τους οικείους και συγγενείς και την ε, ε, ε, ένωση, επανένωση οικογενειών και την προστασία έναντι απελάσεων. Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να υπαγρυπνήσουμε ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου, ώστε οι κανόνες περιελευθερίας κυκλοφορίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σεβαστοί. Και όταν πρόκειται για εκλογικά δικαιώματα πάλι έχουμε εντοπίσει στην έκθεση για την ηθαγένεια και τα δικαιώματα των πολιτών και στην έκθεση όσον αφορά για τις ευρωεκλογές ε, που, έκθεση που εγκρίθηκε έχουμε εντοπίσει θέματα που αποτελούν προσκόμματα και παρακολύουν τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων τους. Για παράδειγμα, όσον αφορά την καταχώρηση ή σε μητρώα ή την απουσία τέτοιων ε, ρυθμίσεων, πώς μπορούν να ασκηθούν αυτά τα δικαιώματα. Έχουμε ξεκινήσει διάλογο με τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη. Αρκετά κράτη-μέλη είπαν ότι θα τροποποιήσουν την νομοθεσία τους και βρισκόμαστε σε επαφή με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη ώστε να διασφαλίσουμε ώστε θα συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε, Έχουμε και το 2013 ως το έτος, Ευρωπαϊκό έτος για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και τα δικαιώματα των πολιτών. Θα δώσει την ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες, τα άτομα, για τα εκλογικά τους δικαιώματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να συζητήσουμε και θα συζητήσουμε και για το ευρωπαϊκό έτος ε, της Ιθαγένειας, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να σας υπενθυμίσω την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, 16 Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης 5 Δεκεμβρίου, έτσι προβλέπετε. Αυτά. 16 λοιπόν του μήνα για τις τροπολογίες κύριος ε, Κύρκοπ έφτασε, οπότε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι η χρησιμοποίηση των προσωπικών στοιχείων επιβατών, PNR. Αυτό είναι το επόμενο σημείο στη μεσιά διάταξη. Ξέρετε ότι το έχουμε συζητήσει στις 13 Ιουλίου. Να σας πενθυμίσω ότι πρόκειται για μια νέα πρόταση μετά την πρόταση του 2007, πριν τη Λισαβόνα, διάφορες απόψεις από διαφορετικούς οργανισμούς, η DPS, η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29, Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έκαναν τις προτάσεις τους και τα βασικά θέματα ήταν το πεδίο εφαρμογή και ο στόχος, οι ορισμοί, η αναλογικότητα, προστασία δεδομένων, η περίοδος ε, της ε, διατήρηση των στοιχείων κτλ. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας κύριο Κύρκο, μετά θα μιλήσουν οι εκπρόσωποι Κομισιών Συμβουλίου και στη συνέχεια θα συζητήσουμε στην Επιτροπή μας. κύριο Κύρκο, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσω, για να σας δώσω τα πιο τελευταία στοιχεία, θα ήθελα να δώσω στην Επιτροπή μας ε, κάποιες ενδεικτικές ε, ημερομηνίες που φαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν είχαμε στη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, αυτό που προτείνω είναι μετά από πολύ επιτυχημένη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο για να δούμε εκεί πώς ε, τα θέματα των δεδομένων και τα ελληνιακά θέματα αντιμετωπίζονται ε, σε ό,τι αφορά το PNR με παρουσία αρκετών συναδέλφων ε, θα ήθελα στις 22 Νοεμβρίου να γίνει μια συνεδρία των σκιωδών συγητών. Εκεί διάφοροι προσκεκλημένοι θα μας ε, παρουσιάσουν την άποψή τους για την επεξεργασία αυτού του συστήματος PNR προσωπικών στοιχείων επιβατών και ίσως μας απαντήσουν και κάποια δύσκολα ερωτήματα που θα τους ε, θέσουμε για το κατά πόσο είναι εφικτό, μάλλον ευκταίο να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα. Και αυτό βέβαια στις 20 Νοεμβρίου. Η έκθεσή μου τώρα θα υποβληθεί, έτσι σκοπεύω, στις 10 Ιανουαρίου και προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών μπορεί να είναι 20 Ιανουαρίου και μπορούμε να ψηφίσουμε το Φεβρουάριο το σχέδιο έκθεση. Σας φαίνεται ότι είναι μακριά ίσως ε, χρονικά, δεν είναι και τόσο όμως, δεν απέχει και πολύ. Άλλωστε πάντοτε θέλαμε ότι στόχος μας είναι να έχουμε μια σωστή πρόταση και όχι να σπεύσουμε και να ε, έχουμε κάτι που δεν θα είναι σωστό. Απλά θα έχουμε τηρήσει κάποια χρονοδιαγράμματα. Θα ήθελα τώρα, κυρία Πρόεδρε, να σας ε, υπενθυμίσω ε, κάποια γενικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε εκ νέου ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πριν από ορισμένες εβδομάδες είχαμε μια αρχική συζήτηση. Έκτοτε έγινε η δεύτερη συνεδρία των σκιωδών εισηγητών και μετά την τελευταία μας συνεδρίαση και χρήσιμες επισκέψεις και συναντήσεις, οποίες ε, συμμετείχα και εγώ προσωπικά για να δούμε τα θέματα τα οποία είχαν θέσει και οι σκιώδεις εισηγητές ε, εκ του σύνεγγης. Θα ήθελα να σας τονίσω εδώ κάποια θέματα τα οποία είναι νομίζω και συστατικά στοιχεία της όλης μας δουλειάς, αλλά αφορούν και κάποιες ανησυχίες που προκύπτουν. Πρώτα απ' όλα, αποκεντρωμένο ή συγκεντρωτικό, κεντρικό σύστημα, ένα ερώτημα. Ίσως κάποιοι θα θεωρούσαν ότι είναι προτιμότερο και ίσως αναγκαίο ένα κεντρικό σύστημα. Αν δούμε το κόστος πολύ προσεκτικά, καθώς και θέματα όπως η θέση, η πολιτική η οποία μπορεί ε, να ε, αρχίσει να αναπτύσσεται γύρω από όλο αυτό το θέμα, ίσως να μην είναι η καλύτερη δυνατή λύση από τις παρούσεις χρονικής στιγμής. Τώρα, η οδηγία, κατευθυντήρια γραμμή, θα παρέχει τα ίδια επίπεδα ασφαλείας, πρότυπα, προστασία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και παρότι το σύστημα δεν θα είναι κεντρικό, θα δημιουργήσει κεντρικά πρότυπα τα οποία θα ε, πρέπει να εφαρμόζονται. Και νομίζω ότι αυτή είναι η βέλτιστη προσέγγιση. Δεύτερον, θα το πω, το έχω ξαναπεί, κάποιοι συνάδελφοι δεν ήταν τόσο σίγουροι, είναι ένα σύστημα όπου η συγκέντρωση έχει να κάνει πιο πολύ με τη συνεργασία παρά με την επιβολή. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια συστήματα προσωπικών στοιχείων επιβατών τα οποία ήδη ισχύουν ή άλλα τα οποία θα εφαρμοστούν σύντομα. Το σημαντικό εδώ είναι να έχουμε πρότυπα που θα επιτρέψουν τη συνεργασία για να έχουμε ένα σύστημα χρήσιμο σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, ε, δεν χρειάζεται καταναγκασμός ή επιβολή. Συνεργασία είναι το σημαντικό κριτήριο εδώ. Είχαμε κάποιες συζητήσεις επίσης ό,τι αφορά τον κατάλογο σοβαρών εγκλημάτων και τι πεδίο εφαρμογή θα έπρεπε να καλύπτει αυτή η πρόταση για τα προσωπικά στοιχεία επιβατών. Σε ό,τι αφορά τα θέματα επίσης της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας έγιναν κάποιες συζητήσεις και θα ήθελα η συζήτηση αυτή να, είναι πιο πολύ για τα τεχνικά ε, στοιχεία και τεχνικές απαιτήσεις και όχι απλά μια ανταλλαγή επιχειρημάτων. Είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε με μία πρόταση να καλύψουμε τα πάντα. Έχουμε μία ένωση με 27 κράτη-μέλη. Διαφορετικές είναι οι ιστορίες ε, των σύγχρονων αυτών κρατών. Μου το έχουν επισημάνει συνάδελφοι και επομένως διαφορετική είναι η έμφαση ανάλογα με το κράτος μέλος ε, για το οποίο εκάστοτε συζητούμε. Άρα μπορούμε να έχουμε το ένα μέγεθος για όλα. Επίσης, η Επιτροπή μας και το ε, Κοινοβούλιο θα πρέπει να βρούμε ένα επίπεδο, ένα χρονοδιάγραμμα που θα μπορούσε να είναι εφικτό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες. Τα δεδομένα είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Το εξετάζουμε επί του παρόντος και σε άλλες οδηγίες. Στην προκειμένη περίπτωση, στην προκειμένη έκθεση, στόχος μου είναι τα δεδομένα να τα αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη προσοχή και ευαισθησία. Και τα δικαιώματα των ατόμων σε ό,τι αφορά τα δεδομένα τους είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να το παραγνωρίσουμε. Πολύ απλό. Και ξεκάθαρο είναι αυτό. και πρέπει να υπάρχει και μια διαδικασία αξιολόγησης και αναθεώρησης. Πρέπει να είναι συνεχής αυτή η αξιολόγηση και επανεξέταση. Και ίσως θα πρέπει και κάποια ζητήματα που αφορούν τα δεδομένα να τροποποιούνται, αν αυτό καταστεί απαραίτητο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα στοιχεία των προσωπικών στοιχείων επιβατών αεροπορικών μεταφορών, ξέρουμε ότι υπάρχουν απεριόριστε διαδρομέ ε, για πτήσει από ε, και προ χωρών μελών τη Ένωση αλλά και εκτό. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κενό ασφαλεία, γιατί ξέρουμε ότι τα αεροδρόμια μα είναι όλο και πιο ε, πολυάσχολα και όλο και πιο ποικίλουν οι, μετα, οι διάφορες διαδρομές, οι διάφορες δυνατότητες. Σίγουρα δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε με μεγαλύτερο κόστος Ιδίω αυτέ τι μέρε που ζούμε σήμερα, ούτε τον Ευρωπαίο φορολογούμενο πρέπει να επιβαρύνουμε, ούτε τι ήδη βεβαρημένε ε, αεροπορικές βιομηχανίε στην Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι κάποια σέντ παραπάνω στο κόστο του εισιτήριου νομίζω ότι είναι μια εύλογη τιμή αν θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία με αυτό το νέο σύστημα. Και επίση θα το τοποθετούσα αυτό και στο πλαίσιο κάποιων άλλων επιβαρύνσεων και χρεώσεων που φαίνεται ότι συνεχώ προστίθενται ε, στα εισιτήρια η αναλογία ε, της τιμής του εισιτηρίου που πηγαίνει στο κόστος αεροδρομίου, ε, στη, στο πετ, ε, στην κυροζήνη κτλ. Όλα αυτά αυξάνονται και τα λίγα σέντ τώρα που, για τα οποία συζητούμε για την ασφάλεια δεν νομίζω ότι είναι και ένα τίμημα τόσο πια σημαντικό. Και ένα τελευταίο σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι πόσο σημαντικό είναι να έχουμε στα χέρια μας ένα αποτελεσματικό εργαλείο επανόρθωση σε ό,τι αφορά πληροφορίες για στοιχεία, προσωπικά στοιχεία επιβατών, redress. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό γιατί αν υπάρξει κακή χρησιμοποίηση κάποιων δεδομένων, αυτό θα πρέπει να καταλήγει σε κάποια ποινή με τον έναν άλλο τρόπο. Ε, κάθε πολίτης θα πρέπει να μπορεί να ξέρει τι γίνεται με τα προσωπικά του δεδομένα και να μπορεί σε περίπτωση που αυτά δεν χρησιμοποιούν τον σωστό τρόπο να ε, προσφύγει για επανόρθωση, για αποκατάσταση. Κάποια κράτη-μέλη έχουν δείξει απροθυμία. Φαντάζομαι τι επόμενε εβδομάδε, τέλο πάντων ελπίζω να μπορέσω να δείξω με βοήθεια από επαγγελματίε και επιστήμονε γιατί είναι αναγκαίο αυτό, γιατί η αναγκαιότητα εντάσσεται στι προσπάθειέ μα. Ελπίζω όμω ε, να υπάρξει κοινό έδαφος, προθυμία μεταξύ των συναδέλφων σχεδόν και να προχωρήσουμε επικοδομητικά και τελικά να καταλήξουμε σε μια συμφωνία καλή και υλοποιήσιμη. Ένα ευρωπαϊκό σύστημα προσωπικών στοιχείων επιβατών θα ήταν πολύ καλό για την καταπολέμηση της διακρατικής διασυνοριακής τρομοκρατίας και εγκληματικότητας. Δεν είναι απάντηση σε όλα, δεν είναι πανάκια σε όλα, αλλά είναι μια σημαντική βοήθεια στην καταπολέμηση του εγκλήματος και αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρούμε δεδομένων των συνθήκων στι οποίε ζούμε αυτή την περίοδο. Επίσης θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν θα αναπτύσσουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες και θα επισερχόμεθα σε λεπτομέρειες πάνω σε αυτά. Πρέπει να ξέρουμε ότι το σύστημα αυτό έχει ως στόχο ε, να ε, βοηθήσει την σύλληψη ε, βιαστών, λαθρεμπόρων, παιδεραστών, εγκληματών, εγκληματιών, όλων αυτών των κατηγοριών που θέλουμε να περιορίσουμε τη δράση τους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη και γίνεται διμερής ανταλλαγή τους. Μήπως καλό θα ήταν αυτό ε, μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και αν ε, δεν πετύχει η έκθεσή μου. Μήπως θα ήταν καλύτερο να είναι σαφέστεροι και ισχυρότεροι κανόνες ό,τι αφορά την εποπτεία ε, για ένα τέτοιο σύστημα και τους τρόπους προσφυγής. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσε να το εμπιστευτεί αυτό το σύστημα και ο κόσμος, αλλά και οι επαγγελματίες, οι αεροπορικές εταιρείες και οι άλλοι επαγγελματίες του κλάδου. Με πολύ ενδιαφέρον και προσοχή θα ακούσω τις απόψεις σας και θέλω να σας ε, διαβεβαιώσω ότι είμαι πρόθυμος να καταλήξουμε σε μια ως το μεγαλύτερη συνένεση για να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Η πρώτη σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την... Ευχαριστώ λοιπόν. Θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αμέσως μετά στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχοντας ακούσει την παρουσίαση την οποία έκανε ο εισηγητής σας, διαπιστώνω ότι υπάρχει <clears throat> πολύ κοινό έδαφος ανάμεσα σε αυτά τα οποία μόλις είπε και στις δικές μας προτάσεις. Με εξαίρεση βέβαια πιθανώς του εάν η οδηγία αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί και σε εσωτερικές πτήσεις. Απόψή μας σε αυτή τη φάση είναι ότι θα προτιμούσαμε να υπάρξει μια πιο σταδιακή εφαρμογή του PNR στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζοντας το σύστημα αυτό στις διεθνείς πτήσεις, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς χώρες εκτός. Κάτι το οποίο δεν θα έχει κανένα ρόλο να παίξει σε σχέση με το αν πηγαίνει σε χώρα Σέγγεν ή όχι. Δύο χρόνια μετά από την θέση σε εφαρμογή της οδηγίας θα γίνει αξιολόγηση για να δούμε αν η ε, ρύθμιση αυτή θα διευρυνθεί και προς τις εσωτερικές πτήσεις. Νομίζω ότι το σκεπτικό και τα επιχειρήματα για την εφαρμογή του συστήματος αυτού στις διεθνείς πτήσεις είναι σαφή. Και γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι μια πιο σταδιακή εφαρμογή είναι η σωστότερη. Θα ήθελα με αφορμή τη συζήτηση αυτή, αν και δεν είναι επίσημα το θέμα σε συζήτηση, να σα ενημερώσω για τις διαπραγματεύσεις για τα PNR ανάμεσα στην Ευρώπη και τι Ηνωμένε Πολιτείε. Θα ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές πάρα πολύ σύντομα. Το κείμενο θα σας αποσταλεί μέσω των γνωστών εμπιστευτικών δικτύων στο τέλος της εβδομάδας. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια συμφωνία στην οποία να καταλήξουμε ήδη στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Δεν μπορώ να σας πω σε αυτή τη φάση περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία, αλλά να σας προκαταλάβω ο λίγων ότι θα υπάρξει μια τέτοια συμφωνία και θα υπάρξει και συζήτηση για το περιεχόμενό της. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Κάκοπ που μας είπε το πώς πηγαίνουν ε, τα στάδια για τα PNR από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά σιγά. Ίσως είναι και ο τέταρτος χρόνος συζητήσεων. Αυτό αποδεικνύει από τη μία ότι τα κράτη-μέλη προσπαθούν να προτείνουν την καλύτερη δυνατή λύση και από την άλλη βέβαια φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα για το πώς θα πρέπει να είναι το σύστημα αυτό και αν πράγματι θέλουμε ένα τέτοιο σύστημα. Εγώ δεν θα ήθελα να πω ότι τα κράτη-μέλη έχουν τις ίδιες ξεκάθαρες απόψεις για όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Όχι, είναι περίπλοκα τα θέματα, είναι σύνθετα, υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες και διαφορετικές απόψεις για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα συγκυριακά προβλήματα και το θέμα της αναλογικότητας. Νομίζω όμως ότι ένα από τα πιο βασικά προβλήματα είναι ότι προς το παρόν μπορούμε να πούμε σαφώς ότι τα κράτη-μέλη σκοπεύουν να καταλήξουν σε μια κοινή αντίληψη η οποία θα επιτρέψει στο σύστημα αυτό να λειτουργήσει και δεν υπάρχει συζήτηση νομίζω πλέον ουσιαστικά για το αν θα υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα ή όχι. Πρέπει να υπάρξει. Το θέμα είναι πώς θα εργαστεί ένα τέτοιο σύστημα στα πλαίσια μιας πραγματιστικής συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Έχουν υπάρξει επαφές και σε επίπεδο διμερών και πολυμερών ε, σχέσεων και νομίζω ότι στο τέλος θα καταλήξουμε και θα συμφωνήσουμε σε ένα κοινό σύνολο κανόνων ανάμεσα στις χώρες και τα όργανα. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θα ήθελα να σας πω το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και ποιος είναι ο στόχος της Πολωνικής Προεδρίας σε σχέση με το κείμενο τουλάχιστον ως παρουσιάζεται τώρα. Θα ακολουθήσουν 12 ή 13 περαιτέρω παρουσιάσεις στα πλαίσια τη ομάδα εργασίας της λεγόμενης του Ζων Βαλ, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρο. Το μέσο αυτό του PNR θεωρείται σαν ένα υγιές μέσο, κάτι το ιδιαίτερα χρήσιμο, και είναι κάτι το οποίο αποδίδει αποτελέσματα στα πλαίσια της καταπολέμησης και πρόληψης μάλλον του οργανωμένου εγκλήματος. Παρ' όλα αυτά, η εμπειρία από τις χώρες που ασχούν ελέγχου στα πλαίσια των PNR μας λέγουν ότι μπορεί να γίνονται οι έλεγχοι αυτοί κάτω από πολύ, μα πολύ συγκεκριμένους κανόνες. Πράγματι συμφωνούμε και εμείς ε, ε, με τη σταδιακή εφαρμογή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτιζόμεθα απόλυτα με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να πω όμως ότι τα κράτη-μέλη και αυτά θεωρούν ότι το σύστημα αυτό χρήζει μιας κάποιας απλούστευσης. Γιατί αν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο τότε η συνεργασία ανάμεσα στις αρχές των κρατών μελών θα είναι ιδιαίτερα βεβαρημένη, περίπλοκη και δύσκολη. Ως εκ τούτου λοιπόν τα κράτη-μέλη σαφέστατα διευκρίνησαν ότι υπάρχει ανάγκη το σύστημα να λειτουργήσει με απλό τρόπο και εδώ έρχονται και κάποιες προτάσεις από πλευράς της Πολωνικής Προεδρίας έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας, να καλύψουμε τις ανάγκες αναλογικότητας, και εδώ νομίζω ότι έχουμε τις ίδιες απόψεις και με τον κύριο Κύρκοπ σε σχέση με τις εσωτερικές πτήσεις. Έτσι λοιπόν το κείμενο του κανονισμού αυτού τελικά να είναι ένα κείμενο απλούστερο από ό,τι υπάρχει σήμερα, τουλάχιστον σε σχέση με τις εφαρμοστικές του πλευρές. Ένα θέμα το οποίο ε, έχουμε διευκρινίσει πλήρως και συμφωνεί και ο εισηγητής είναι το θέμα της αναθεώρησης της δυνατότητας ανταλλαγής ε, πληροφοριών, εμπειριών, συναντήσεων, μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων κατά κάποιο τρόπο, οι οποίοι θα μπορούν σε μόνιμη, σε ουσιαστικά μόνιμη βάση να ανταλλάσσουν εμπειρίες για να γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει, πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Αυτό είναι το κάτι το πολύ θετικό και θα βοηθήσει ιδιαίτερα τη σωστή λειτουργία του συστήματος. Στα πλαίσια της ομάδας εργασίας Val μιλήσαμε και για το θέμα του κόστους. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς σε σχέση και με τις οικονομικές ανάγκες της ε, ύπαρξης και λειτουργίας των ομάδων αυτών για τα στοιχεία των επιβατών. Τι θα κοστίσει η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος και για τα κράτη-μέλη, τις τους και για τις αεροπορικές εταιρείες. Εν πάση περιπτώσει είμαι στη διάθεση όλων των μελών από εδώ και πέρα. Θα είμαι σε συνεχή επαφή με τους συναδέλφους που ασχολούνται με το θέμα και με τον εισηγητή τον κύριο Κέρκοπφ είναι κάτι το οποίο αφορά και ενδιαφέρει και την Πολωνική Προεδρία και την επερχόμενη Δανική Προεδρία. Ελπίζω να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστούμε. Σίγουρα θα μπορέσουμε, ελπίζουμε, να κινηθούμε σε αυτά τα κοινά θεμέλια αγοργά. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και έτσι θα έχουμε χρόνο για συζήτηση. Άλμπρεχτ παρακαλώ πρώτα. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, Κάπως εκπλήσωμε πρέπει να πω για την ταχύτητα με την οποία προχωρούμε εδώ. Μια και έχουμε διαφορές που βρίσκονται στο τραπέζι και απορρέουν. Το βρίσκω θαραλέο. Με την αποθήκευση δεδομένων και τις επικρίσεις που ασκήθηκαν όσον αφορά την αξιολόγηση αυτών των στοιχείων, των αποθηκευμένων στοιχείων και όσον αφορά και τις ε, τηλεπικοινωνίες και μέσω των συνταγματικών δικαστηρίων των κρατών μελών που ασκήθηκε επίκριση σε αυτή την αποθήκευση, προσωπικών δεδομένων αποθήκευση και βρίσκεται επί τραπέζης παρόλα αυτά το θέμα. Το βρίσκω λοιπόν θαραλέο πώς το προσεγγίζουμε. Τώρα, σε σχέση με τις αρχές των συνταγμάτων των κρατών μελών, αυτό δεν είναι, θα έλεγα, δεν συνάδει και με την Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε και με το άρθρο 16 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρίσκω θαραλέο όμως γενναίο, επειδή η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου αυτές τις επικρίσεις και αυτή τη συνταγματική κατάσταση και τις επικρίσεις και επιφυλάξεις ε, ανέφερε και τα υπέβαλε στο Συμβούλιο και είναι γνωστό ότι υπάρχουν αυτές οι επικρίσεις στο Συμβούλιο. Είναι ακόμα πιο θαραλέο ότι η υπηρεσία δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ότι ο υπεύθυνο ε, για τα ε, προσωπικά δεδομένα άσκησαν τέτοιε επικρίσεις για την αποθήκευση για πενταετή περίοδο και παραπάνω που δεν είναι καθόλου αναλογική υπόθεση και μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αποδείξεις για την αναγκαιότητα αυτής της χρονικής διάρκειας αποθήκευσης. Το βρίσκω γενναίο και θαραλέο επειδή οι εταιρείε εναέριων μεταφορών, οι carriers, έχουν επισημάνει ποιο κόστος θα συνεπάγεται αυτό. Η Lufthansa και μόνο είπε ότι για αυτή την πρόταση που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι 200.000 ευρώ ε, κάθε μήνα πρέπει να δαπανώνται. Αν πάρουμε και τις πτήσεις όπως αναφέρει τώρα τις, ε, οι ευρωπαϊκές θα πάμε στα εκατομμύρια όπως προτείνει να γίνεται ο κύριος Κέρκοπ σε οικονομική κρίση και συγκυρία χρηματοοικονομικών περικοπών και λιτότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα εισαγάγουμε ένα σύστημα το οποίο θα προκαλέσει τεράστιες δαπάνες για τους φορολογούμενους ή για τους Ευρωπαίους πολίτες και καταναλωτές. Τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος τέλος είναι απίστευτο ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν καν αποδείξεις ότι είναι αναγκαία όλα αυτά και υπάρχουν κριτικές παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί και παρόλα αυτά συνεχίζουμε σαν να μην υπάρχει τίποτα ως επιφύλαξη. Δεν το κατανοώ πλέον, είναι ασύλληπτο, δεν το καταλαβαίνω και αυτή την πρόταση δεν μπορώ να την υποστηρίξω καθόλου. Και θέλω να καταστήσω σαφές ότι είμαι ένας από εκείνους εγώ που εννοούσε προσωπικά ο κύριος Κέρκοπ, ότι έχουν λέει μεγάλες αμφιβολίες αν ένα τέτοιο σύστημα είναι αναγκαίο. Σωστό, δεν είναι αναγκαίο και επικεντρωνόμαστε σε άλλα είδη ε, ε, αστυνομικής συνεργασίας και όχι τη συλλογή και αποθήκευση όλων των ατόμων και των προσωπικών τους δεδομένων που θα αναλύονται διαρκώς και θα υπάρχει μια διαρκής αστυνόμευση και θα πρέπει εδώ να αποδεικνύει κανείς πάντα ότι είναι αθώος όχι να αποδεικνύεται ότι είναι ένοχος αλλά να αποδεικνύεται διαρκώς ότι κάποιος είναι αθώος αυτά είναι ασύλληπτα πράγματα και ότι όταν κάποιος μεταφέρει υπερβολικά πολλές αποσκευές ε, ή έχει κάποιο λάθος όνομα με το οποίο καταχωρήθηκε ή έχει κάποιες επιθυμίες για τα γεύματά του στα αεροπλάνα, ε, δεν είναι δυνατόν η αστυνομική συνεργασία εκεί να, να επικεντρώνεται. Πρέπει να υπάρχει μια βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των αστυνομικών αρχών και των ε, κυβερνήσεων και αρχών των κρατών μελών. Σωστό, αναγκαίο αυτό. Όμως αναγκαία στοιχεία και όχι περιτά και σίγουρα να δούμε τι πρέπει να αποθηκεύεται. Αλλά αποθήκευση συλλήβδην προσωπικών δεδομένων αθώων ανθρώπων που δεν είναι ύποπτοι όλων των πολιτών και που ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό δεν είναι αναλογικό, δεν είναι λογικό και δεν είναι ισοβαρές και δεν συνάδει με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν και ιδιαίτερα υπέρμαχος ενός συστήματος προσωπικών στοιχείων επιβατών. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το γενικό ζήτημα, αυτό της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και γνωρίζουμε ότι έχει ε, προειδοποιήσει η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου την Κομισιόν και κατ' επέκταση και εμάς τελικά ε, σε ό,τι αφορά την πρόταση αυτή που πρέπει να συνάδει με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Επίσης κάποιοι από εμάς δεν είμαστε βέβαιοι ότι το 100% του χρόνου κάνουν τα κράτη-μέλη ό,τι είναι δυνατόν και εφικτό για να αποφύγουν γνωστή υποπτή, γνωστή ε, τρομοκράτες, εγκληματίες τέλο πάντων άτομα για, για τα οποία υπάρχουν στοιχεία ότι θα μπουν ε, στη χώρα, είτε μέσω κάποιων ε, ελέγχων πολύ ενδελεχών στα σύνορα ή με κάποιες λίστες. Τέλο πάντων υπάρχει ιδιαίτερη αμφισβήτηση και στη χώρα με όλα αυτά τα θέματα. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι έχουν γίνει όλα όσα είναι αναγκαία για να σταματήσουμε αυτά τα άτομα. Και αυτό έχει να κάνει με όλων των ειδών συλλογής δεδομένων και τέτοια προγράμματα. Αυτή είναι η μία ανησυχία και η δεύτερη είναι ανησυχίες για την ασφάλεια των δεδομένων, να σταματήσουμε την μη εξουσιοδοτημένη παράνομη χρήση δεδομένων. Και υπάρχει και η κοινοποίηση ε, ασφαλείας που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Το Security Breach Notification. Έχουμε κάποιες διατάξεις στη συμφωνία με την Αυστραλία για ένα σύστημα προσωπικών στοιχείων επιβατών ε, Αυστραλίας για την εξατομίκευση των στοιχείων και της καταγραφής για να υπάρχει ασφάλεια των στοιχείων και προστασία του. Ειδικά σε ό,τι αφορά το PNR τώρα. Αυτό που πάντοτε με ανησυχεί και με ανησυχούσε ήταν το profiling των ε, χρηστών. σαν χαλασμένο γραμμόφωνο είμαι. Ίσως τέλο πάντων επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δέχεται να χρησιμοποιήσει αυτόν τον, τον ε, όρο profiling, είτε στην πρόταση είτε στο οπουδήποτε αλλού. Νομίζει ότι εφαρμόζεται μόνο στην αυτόματη λήψη αποφάσεων ε, για να μην μπει κάποιος ε, στο έδαφος μιας χώρας. Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι σημαίνει αυτό. Αν δει κανεί ε, την, την επεξηγηματική, την ιδεολογική έκθεση της Κομισιόν, θα δει ότι λέμε, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε πραγματικό Χρόνο βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων για να καθοριστεί κατά πόσον κάποια άτομα θα πρέπει να ελεγχονται. Οι λεγόμενοι άγνωστοι ύποπτοι να καλύπτονται από αυτό. Τώρα ύποπτοι άγνωστοι δεν υπάρχουν. Γνωστοί μόνο είναι. Και αν θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο, ας πείτε τα πράγματα με το όνομά του. και ας πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν απαραίτητε ασφαλιστικές δικλείδε. Δεν νομίζω ότι βοηθάει να το γυρίζουμε γύρω-γύρω και να μην το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Ουσιαστικά τι θέλουμε να φτιάξουμε, ένα στερεότυπο, ένα παράδειγμα των ατόμων για τα, τα οποία πρέπει να ελέγξουμε. και δημιουργούνται κάποια κριτήρια αξιολόγηση. Εγώ θα το έλεγα profiling αυτό, δημιουργία προφίλ. Και αυτό θα το εφαρμόσουμε σε κάποιε πτήσει ή σε πτήσει από ένα συγκεκριμένο προορισμό. Ωραία. Και υπάρχουν λοιπόν τότε κάποια άτομα τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέταση. Αυτό θα προκύψει με όλη αυτή την ανάλυση. Εντάξει, μέχρι ένα σημείο όμω. Δεν είναι το θέμα αν θα μπουν για δευτερεύοντα έλεγχο κάποια άτομα, αλλά Αυτά τα στοιχεία διαγράφονται από το σύστημα μετά. Δηλαδή, εάν αποφασιστεί ότι μετά την έρευνα δεν ε, ε, περαιτέρου ανάλυση σε ένα άτομο, τι γίνεται με αυτά τα στοιχεία, διαγράφονται. Γιατί με αυτούς τους μη γνωστούς υπόπτους το πρόβλημα είναι ότι πρέπει κανείς να αποδεικνύει ότι είναι αθώος, μεν, αναστροφή βάρους απόδειξης, άρα ένα βάρος αυτό, αλλά η παράδοση γι' αυτό γινόταν ε, το λεγόμενο rendition. Δηλαδή βρίσκαμε κάποια άτομα τα οποία ήταν σε λάθος χρόνο τη λάθος στιγμή. Κάποια από αυτά τα άτομα μπορεί να ήταν ένοχα, μπορεί να μην ήταν όμως κάποια άλλα για τίποτα ένοχη. Απλά τέριασαν σε ένα προφίλ αυτό ήταν το πρόβλημα. Και όλα, όλοι γνωρίζουμε που μπορεί να καταλήξει αυτό. Αυτό που θέλω εγώ να φροντίσουμε είναι τίποτα φρικτό, άβολο, ανήσυχο. Άτομα τα οποία έχουν επισημανθεί μέσω αυτού του profiling, γιατί πρέπει να το δεχθεί η Κομισιόν ότι περί αυτού πρόκειται, δημιουργούνται προφίλ θα υπάρχουν διασφαλίσεις ότι κάθε ίχνος, όχι μόνο η ανωνυμοποίηση των δεδομένων, δεν αρκεί αυτό. Όποιοι έχουν περάσει ένα δεύτερο έλεγχο ή κάπως επισημαίνονται ότι πρέπει να ελεγχθούν γιατί μπορεί να χρησιμοποίησαν τον ίδιο ταξιτικό πράκτορα ή να εκδόθηκαν οι κάρτες τους από τον ίδιο κτλ να μην του συμβεί κάτι κακό κάποια στιγμή στην όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό πρέπει να το ε, φροντίσουμε. Τέτοιε διασφαλίσει δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμή γιατί η Κομισιόν δεν κατονομάζει τα πράγματα. Thank you very much, Romero. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ρομέρο παρακαλώ. <clears throat> Ευχαριστώ. Πραγματικά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο θέμα, Πρόεδρε. Δεν πρόκειται για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε έρευνες όσον αφορά εγκλήματα μόνο. Υπάρχει πραγματικά αυτή η συνεργασία στην Ευρώπη και γι' αυτό δημιουργήθηκε η Ευρωπόλ και γι' αυτό δημιουργήθηκε και η Eurojust. Το πρόβλημα είναι ότι ο συντονισμός ακόμα έχει μεγάλες ελλείψεις <clears throat> και αν έχει ελλείψεις ο συντονισμός όταν πρόκειται για έρευνες για ένα έγκλημα και για την εκδίκασή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ταυτόχρονα που στοχεύει, θέλει να δημιουργήσει ένα συντονισμό που ακόμα ωστόσο όμως δεν γνωρίζουμε αν θα είναι εφικτό και δυνατό ή όχι. Αυτά όσον αφορά τις μονάδες πληροφόρησης θα συντονίζουν στοιχεία και προσωπικά δεδομένα ή τι θα κάνουν. Ουσιαστικά πρόκειται για την ίδια την φιλοσοφία της πρόληψης και πρέπει να προβληματιστούμε και να σκεφτούμε και για αυτά τα θέματα. Δεν επιτρέπονται όλα για την πρόληψη εγκλημάτων, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Λοιπόν, οι παράνομες ακροάσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων για παράδειγμα, ε, δεν είναι κάτι το νόμιμο, δεν επιτρέπονται όλα για να γίνονται έρευνες και για να προσάγονται στη δικαιοσύνη κάποιοι εγκληματίες και για τους ταξιδιώτες γνωρίζοντας ότι ε, εδώ πρόκειται να υπάρξει έρευνα των πάντων, τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα είδος, πώς να το πω, προδοσίας των ίδιων των πολιτών από πλευράς μας με τέτοια μέτρα. Δηλαδή γίνεται ύποπτος ο πολίτης εξορισμού και πρέπει να αποδεικνύει ο πολίτης ότι είναι αθώος αντί να αποδεικνύουν οι άλλοι ότι είναι ένοχος. Και όταν πρόκειται για κάποιο σφάλμα τη ίδια τη διοίκηση, πρέπει να λειτουργήσει ένα ολόκληρο μηχανισμό για να μπορέσει να υπερασπίσει τα δικαιώματά του αυτό ο πολίτη. Και όλα αυτά σε σχέση με το μηχανισμό τη πρόληψη. Αυτό ο μηχανισμό τη πρόληψη εισήχθη, διότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει η δυνατότητα με του αναλυτέ των αστυνομικών αρχών να έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε εκατομμύρια εκατομμυρίων προσωπικών δεδομένων. Τεχνολογικά, από πλευρά τεχνική και τεχνολογία, αυτό είναι εφικτό. Το γεγονό ότι αυτό είναι εφικτό και δυνατό, τι σημαίνει. Ότι δεν θα αξιολογήσουμε εμεί ποια είναι τα όρια όλων αυτών των πράξεων. Γιατί θα πρέπει, πρέπει να αξιολογήσουμε ποια είναι τα όρια αυτού του επίπεδου πρόληψης. Ίσως όταν του λένε κάποιου ταξιδιώτη ότι χάρη σε αυτές τις δράσεις μπορεί να, μην, να αποφευθεί μια βομβιστική απόπειρα σε ένα ε, αεροπλάνο εντάξει μπορούμε να κάτι τέτοιο να το δεχθούμε ως ε, ε, ανακούφιση το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν έχουν καθοριστεί αυτά εξειδικευμένα όταν γίνεται λόγο για σοβαρά εγκλήματα και παραπτώματα υπάρχει ένα πολύ ευρύ πεδίο εφαρμογής και ουσιαστικά όσον αφορά τις μονάδες ε, πληροφόρησης δεν είναι μόνο για πληροφόρηση και έλεγχο των στοιχείων. Είναι επίσης αυτές οι μονάδες, μονάδες έρευνας και ανάκρισης και δικαστικών ε, κρίσεων και αποφάσεων. Πώς μπορούν όλα αυτά να γίνονται και ε, σε σχέση με αυτά τα πλαίσια. Είναι προφανώς αστυνομικές μονάδες και δικαστικές μονάδες Ποια σχέση έχουν αυτές οι μονάδες τώρα με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Γίνεται λόγος στην οδηγία για αυτά τα πράγματα, αλλά δεν καθορίζονται με κανένα τρόπο πώς θα γίνονται όλα αυτά. Όταν έχουμε δικαστική και αστυνομική ε, τέτοιου είδους δράση, πώς θα γίνεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όλα αυτά χωρίς να έχουν καθοριστεί, χωρίς να υπάρχουν όρια και σαφείς γραμμές. Πρέπει λοιπόν να προβληματιστούμε και να σκεφτούμε τι θα γίνει σε αυτό το επίπεδο. Ακόμα και στο επίπεδο των κυρώσεων δεν υπάρχει σαφήνεια. Είναι σαφέ. οι κυρώσει και τα πρόστιμα και οι ποινέ είναι πολύ διαφορετικές σε σχέση με τα κράτη μα. Κάθε κράτος θεωρεί ότι εδώ βλέπουμε ότι ξεπερνάμε σαφώς κάποια όρια. Υπερβαίνονται τα όρια της, ε, των εγγυήσεων του κράτους δικαίου. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα έκτακτο, ξεχωριστό μέσο εδώ, ειδικό μέσο και πρέπει να προβληματιστούμε σε βάθος να δούμε τι θα γίνει για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων. Να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο και καταλήξουμε στο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός τρευλός που δεν θα προστατεύει τους πολίτες και δεν θα πρέπει κιόλας και να χρησιμοποιείται. Τι είδους εχέγγυα θα υπάρχουν, τι είδους ε, δράσεις για το πεδίο εφαρμογής θα υπάρχουν. Ποια περίοδος χρονική για την αποθήκευση και παρακράτηση στοιχείων θα προβλέπετε. Όλα αυτά πρέπει να καθοριστούν για να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο σαφές πλαίσιο. Ε, ευχαριστώ. Νομίζω ο κύριος Γράντες Πασκουάλ είναι επόμενος. Ο μιλητής, ναι, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στην Επιτροπή Μεταφορών για αυτό το θέμα θα γνωμοδοτήσουμε, θα συντάξουμε μια γνωμοδότηση για τα προσωπικά στοιχεία επιβατών και θα ήθελα να σας πω κάποιες σκέψεις. Δεν υπήρξε συνασπισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ Επιτροπής ΛΥΠ, Επιτροπής ε, Μεταφορών. Νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι σαφέ ότι δική σα είναι καταλληλότερη επιτροπή για να αντιμετωπίσει αυτό το λεπτό ευαίσθητο θέμα που αφορά θεμελιώδη δικαιώματα. Εγώ λοιπόν ε, από την ε, θέση μου, από την ιδιότητά μου ως μέλος Επιτροπής Μεταφορών θα είμαι υπέρ του εμείς στην Επιτροπή Μεταφορών να δούμε μόνο τα θέματα που άπτονται ειδικά του τομέα των μεταφορών και δική σας να είναι η ε, Επιτροπή που είναι και η κατεξοχήν ε, αρμόδια και θεματοφύλακα των θεμελιωδών δικαιωμάτων που θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Τώρα, ακούσαμε ουσιαστικά από κάποιους ε, εισηγητέ, από κάποιους ομιλητέ, να μην θεωρούν ότι είναι σκόπιμη η χρησιμοποίηση αυτών των ε, προσωπικών στοιχείων και είπαν ότι χρειάζεται σθένος. Ε, μάλιστα είπαν κάποιοι ότι είναι πολύ ρηψοκίνδυνη και τολμηρή η Κομισιόν όταν προτείνει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι είναι υποχρέωση της Κομισιόν να υποβάλει αυτό το θέμα και στην Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών να το θέσει. Το θέμα της αναλογικότητας μεταξύ του μέσου που χρησιμοποιείται και του στόχου που είναι η καταπολέμηση στην προκειμένη περίπτωση της τρομοκρατίας και η αποτροπή άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Αυτό είναι το θέμα. Αν εμείς στην Επιτροπή μπορούμε να βρούμε την ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο, νομίζω ότι ήδη θα πετύχουμε το στόχο μας. Αν δεν τα καταφέρουμε, τότε θα κάνουμε κάποια υπερβολή. Ίσως θα ε, είναι αυτό το αποτέλεσμα. Είπα ότι η Επιτροπή σα είναι ιδανική ιδανική για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας πάντα υπάρχει ένα λεπτό ζήτημα. Μία διχοτομία ε, μεταξύ ασφάλεια, αφενό, αφενός ελευθερίας αφετέρου. Είναι ένα όριο που δεν μπορεί να το ξεπεράσει κάποιο, Αλλά είναι και ένα μονοπάτι που πρέπει κανείς να το περπατήσει. Και θα πρέπει βέβαια να το κάνει χρησιμοποιώντας όλα τα δημοκρατικά εργαλεία και μέσα για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την τρομοκρατία. Αυτό είναι το, το σημείο κλειδί. Χωρίς δηλαδή υπερβολές να καταφέρουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο στον αγώνα για την ε, καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ίσως αντιμετωπίσουμε προβλήματα ε, ερχόμενοι ε, αντιμέτωποι με κάποιες ευαισθησίες. Ε, η τρομοκρατία, τα σοβαρά εγκλήματα ε, μπορούν να μας δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα στο πώς ορίζονται ή μπορούν να μας δημιουργήσουν πρόβλημα ε, σε κάποια σε νούμερους σε κάποιες ποσοστώσεις. Δεν θα πρέπει να βρούμε παραθυράκια που θα οδηγήσουν σε υπερβολή. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, αλλά το των θέλω να σας πω ότι εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς ε, να απαξιώσει αυτή την πρόταση της Κομισιού γιατί πράγματι πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το ζήτημα. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας απαιτεί αποτελεσματικά εργαλεία. Δεν είναι ε, κάτι που είναι από κύμα φαντασίας, τρομοκρατία. Είναι μια πραγματικότητα και θα πρέπει να προστατευτούν από τη τρομοκρατία οι δημοκρατικές κοινωνίες αλλά να το κάνουν με δημοκρατικούς ε, τρόπους και μέσα. Να προστατεύσουν την δημοκρατία. Δεν θα πρέπει αυτά τα εχέγγυα αυτές τις ασφαλιστικές ε, δικλίδες να, βέβαια να τις ε, ε, ξεχνάμε. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Βλέπουμε να υπάρχουν όλο και περισσότερες ανεπάρκειες και όλο και μεγαλύτερα κενά. Νομίζω ότι σε σωστό δρόμο βρισκόμαστε και ο εισηγητής θα κάνει καλή δουλειά. Θα δούμε και με τις τροπολογίες, θα δούμε πώς εμείς μπορούμε αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε από την Επιτροπή Μεταφορών να κάνουμε εδώ στην Επιτροπή σα, σε συνεργασία βέβαια με τον εισηγητή που θα μα δώσει την κατεύθυνση. Εγώ είμαι ένα πληρωματικό μέλο τη Επιτροπή σα, αλλά ε, συζητάω και ασχολούμαι με αυτά τα θέματα και στην Επιτροπή Μεταφορών και θα συνεχίσω να το κάνω. Θα έχουμε μια ήρεμη συζήτηση, συνεργασία, διάλογο για να βρούμε την ισορροπία. Δηλαδή, και να εγγυηθούμε την ε, ασφάλεια αλλά και να διατηρήσουμε την ελευθερία. Θα πρέπει να έχει κάθε κράτος μηχανισμούς για να μπορεί να εγγυάται τις ελευθερίες του. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ε, από ό,τι βλέπω, ε, είναι αρκετά διαφορετικές ε, και αντικρουόμενες οι απόψεις για το θέμα της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας, για το κατά πόσον είναι ανάγκη να υπάρχει εικονισμός ή όχι, για το τα κτλ. Θα ζητήσω από την Κομισιόν πρώτα να μας δώσει τις δικές της σκέψεις πάνω σε όλα αυτά και εν συνεχεία στο Συμβούλιο αν θέλει να λάβει το λόγο. Κομισιόν λοιπόν και μετά ο κύριος Κύρκοπ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια από τα θέματα και παρατηρήσεις που έγιναν εδώ. Όσον αφορά την θέση του Συμβουλίου, της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου, θεωρούμε ότι πρόκειται μάλλον για μια μάλλον αντινομοθετική πρόταση παρά νομοθετική γνώμη, νομική γνωμοδότηση. Παρ' όλα αυτά δεν θα αποφύγω να συζητήσω και να προσεγγίσω το θέμα της εναλλακτική νομικής πρότασης ως εξή. Υπάρχει η θελκτική ιδέα των targeted flights, στοχοθετημένων πτήσεων, λέγοντας ότι μόνο για αυτές τις στοχοθετημένες πτήσεις θα εφαρμόζεται αυτή η διάταξη, θα εφαρμόζονται αυτές τις διατάξεις και για τις επικίνδυνες διαδρομές. Δεν νομίζουμε ότι κάτι τέτοιο όμως μπορεί να λειτουργήσει. Θα σας πω γιατί διότι έχουμε κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχουν δικαιώματα να γνωρίζουν οι πολίτες ποιες είναι οι στοχοθετημένες διαδρομές. Και αν υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα για αυτές τι στοχοθετημένες διαδρομές και υπάρχουν κάποιοι εγκληματίες ή θέλουν να κάνουν κάποιες εγκληματικές πράξεις, θα αποφύγουν αυτές τις ε, επικίνδυνες διαδρομές χρησιμοποιώντας κάποιες άλλες εναλλακτικέ διαδρομές. Νομίζουμε ότι είναι πολύ εύκολο λοιπόν να παρακαμφθεί αυτό και αυτό θα οδηγήσει σε κάποια υποκριτική αντιμετώπιση αν δεν ληφθεί αυτό υπόψη. Θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα εφαρμόζεται για όλες οι λίβδιν της πτήσης διότι όλες οι πτήσεις θα είναι εναλλακτικέ δυνάμει διαδρομές έναντι των επικίνδυνων πτήσεων. Ή θα έχουμε κάποιες εναλλακτικέ διαδρομές, να δώσουμε την εντύπωση, δηλαδή κάνουμε πολλά για να ενισχυθεί η ασφάλεια. Όμως πάλι μπορεί να παρακαμφθεί κάτι τέτοιο, διότι τρομοκράτες ή εγκληματίες μπορούν και αυτοί να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικέ διαδρομές, έτσι δεν είναι. Πιστεύουμε λοιπόν ότι δεν θα ήταν λειτουργικά όλα αυτά, δεν θα είχαν αποτέλεσμα στο τέλος τέλος. Και κάτι άλλο. Για το κόστος και τα συνολικά στοιχεία. Μπορεί να φαίνεται ίσως εντυπωσιακό, αλλά πρέπει να κάνουμε λόγο ότι κάνουμε λόγο για 0,10 σέντ εισιτήριο και αυτό δεν πιστεύω ότι είναι εκείνο το οποίο θα παρακολύσει την ευρωπαϊκή οικονομία από το να ανακάμψει στο μέλλον. Δεν θα είναι αυτό κάποιο τρομερό, κάποια τρομερή επιβάρυνση. Αν μπορείτε να συντομεύσετε παρακαλώ. Τρίτον, λοιπόν, για το θέμα της ασφάλειας. Σημείωσα τις παρατηρήσεις που έγιναν από την Βαρονέσα Λάτφορντ και θα ήθελα να τη διασφαλίσω να της πω ότι για τα θέματα των, της οδηγίας ε, ε, είναι ισχυρότερα αυτά από την συμφωνία με την Αυστραλία, αλλά με ευχαρίστηση διμερώς να το αποσαφηνίσουμε ή να αυξηθεί το θέμα για την ασφάλεια δεδομένων. Πιστεύουμε όμως ότι είναι αυστηρότερες οι διατάξεις για τις διαδρομές αυτές που έχουμε προβλέψει από ό,τι σε σχέση με τη συμφωνία με την Αυστραλία. Για το θέμα των αξιολογήσεων τάσεων, trend assessment, και το να μην διατηρούνται αποθηκευμένα τα στοιχεία τα οποία εσφαλμένα ίσως μπορούν να κατηγορήσουν κάποιον επειδή βρισκόταν δίπλα σε κάποιον ή χρησιμοποιήθηκε μια πιστοτική κάρτα από το ίδιο ε, ταξιδιωτικό γραφείο κτλ. Τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Εξετάζουμε ευμενώς αυτά τα οποία αναφέρατε. Θεωρούμε ότι έχετε απόλυτο δίκιο στο ότι αυτού του είδους τα στοιχεία θα πρέπει αμέσως να διαγράφονται ή τουλάχιστον ταχύτατα να απορρίπτονται και να διαγράφονται. Και αφορά αυτό τα επιχειρήματα που ακούστηκαν, ότι σε σχέση με τέτοιου, τέτοιου είδους ε, ε, λάθος υποψίες, ε, εσφαλμένες υποψίες πρέπει να αποφεύγονται στο μέλλον. Αλλά με θετικό πνεύμα αντιμετωπίζουμε την πρότασή σας. Ευμενώς αντιμετωπίζουμε την πρότασή σας, ευνοϊκά την αντιμετωπίζουμε μια τέτοια προσέγγιση. Στη συνέχεια τέλος, για να ολοκληρώσω, σημειώσαμε καλώς επίσης αυτά που είπε η κυρία Κάμερο Μέρο. Πιστεύουμε σίγουρα ότι η πρόταση έχει αρκετά ισχυρές αναφορές για την προστασία προσωπικών δεδομένων και όσον αφορά και τις ποινές ή τις κυρώσεις, Ευχαριστώ να επεξηγήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες ε, τι μπορεί να γίνει για να ενισχυθεί αυτή η συνιστόσα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ όπως άκουσα. Υπήρξαν, κάποιε ε, κάποιες, παρατηρήσεις ε, από πλευράς κυρίου Κερκόπ. Εσείς, νομίζω όλοι σας, συγγνώμη πρόεδρε, κάνουμε λόγο σε αυτή τη συζήτηση σήμερα για τη δική μου έκθεση, έτσι, την οποία δεν έχω ακόμα συντάξει. Όλοι καταλήγουν σε συμπεράσματα με βάση αποκλειστικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν έχουμε μια συζήτηση απόψε για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τότε δεν έχει νόημα να παρίσταμε. Εγώ είμαι ο εισηγητής ο οποίος θα υποβάλει την έκθεση, την οποία δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει και συντάξει, για να ακούσω σχόλια και παρατηρήσεις από αυτόν που ανέφερα προκαταρκτικά πριν από τη σύνταξη τη εκθεσή μου. Θα ήμουν ευγνώμων αν τηρούσαμε συζήτηση σε αυτό το περιορισμένο, σε αυτό το περιορισμένο εύρο και όχι επί παντό του επιστητού επί των προτάσεων τη Επιτροπή. Θα προτιμούσα να μην έχουμε ξεχωριστή συζήτηση μεταξύ των συναδέλφων μου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι αυτό το νόημα αυτού του εγχειρήματο. Δεν μα πήγαινε πουθενά. Η έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής έχει υποβληθεί εδώ και αρκετό καιρό. Εμεί έχουμε προχωρήσει προς τα εμπρό. Θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσαμε να περιοριστούμε στη συζήτηση των θεμάτων που είναι υποσυζήτηση όσον αφορά τη δική μου έκθεση. Ευχαριστώ. Δηλαδή, εσείς θα συντάξετε την έκθεσή σας και τότε μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι και να καταθέσουμε να υποβάλουμε τροπολογίες και καθότι γνωρίζουμε η έκθεση δεν θα είναι καθόλου εύκολο εγχείρημα υπάρχουν αντικρουόμενες και αντιφατικές απόψεις, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και τοποθετήσεις. Από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακούγοντας τα όσα ανέφερε ο κύριος Κέρχοπ σε σχέση με τα σχέδιά του και τις απόψεις του για την έκθεσή του, να ληφθούν υπόψη. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση εδώ για αυτό το θέμα απόψε. Το Συμβούλιο όμως ακόμα θα παρέμβει, έτσι. Ε, δεν έχω ολοκληρώσει την παρέμβασή μου, Πρόεδρε, λυπούμε. Τώρα θα έχουμε και το Συμβούλιο. Αλλά, ναι, αλλά η ένδειξη είναι η επισήμαση, όχι σε σχέση με το ότι δεν θα έπρεπε να λυθεί αυτό υπόψη, αλλά να παρέμβει το Συμβούλιο απλώς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε σχέση με τον κύριο Κέρκοπ, μπορώ ουσιαστικά να ανταποκριθώ σε αυτό το οποίο πρότεινε να τοποθετηθώ επ' αυτού. Τολμώ να πω ότι πολύ συχνά θα μπορούσαμε ίσως να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις και προκατηλημένες απόψεις σε σχέση με αυτό το μέσο, το εργαλείο αυτό. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο ε, σε σχέση με την εμπλοκή του κυρίου Κέρκοπ που θα πρέπει να μπορέσει να ε, λάβει υπόψη χειροπιαστά και συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται στη δράση εκείνων που ασχολούνται με το PNR για να δούμε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Εγώ ίδιος επί αρκετό χρονικό διάστημα, έχοντας δει τις αρχικές διατυπώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για όλα αυτά, όχι εξεπλάγιν, αλλά με έκπληξη είδα πόσο αυστηρές προϋποθέσεις εφαρμόζονται και ποια δυνατότητα υπάρχει για κατάχρηση των στοιχείων που είναι πολύ περιορισμένη σε εύρος και γι' αυτό επικεντρωθήκαμε στο έργο αυτής της ομάδας ε, για την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων και σε σχέση με την παρατήρηση για την παραβίαση κάποιων ε, ε, παραμέτρων λαμβάνουμε ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη αυτά τα θέματα και συμμεριζόμαστε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θέλουμε να πάμε και να προχωρήσουμε πολύ πιο πέρα σε σχέση με τη συμφωνία με την Αυστραλία. Θα πρέπει να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο και να είναι ιδιαίτερα απαιτητικέ οι προδιαγραφές και οι ρυθμίσεις. Και τώρα, δεν είμαι σε θέση να ερμηνεύσω σε σχέση με τη, ε, τη γνωμοδότηση από πλευράς της υπηρεσίας του Συμβουλίου. Όμως, όσον αφορά την ε, προσπάθεια που έγινε από πλευράς της ομάδας ήταν η προσπάθεια να ε, ληφθεί υπόψη ότι όταν αναφέρθηκε από την ε, νομική γνωμοδότηση του Συμβουλίου ότι θα έπρεπε να ληφθούν όλες αυτές οι συνιστώσεις υπόψη, αυτό δεν θα συνέβαινε πάντα. Δεν θα είμαστε πάντα σε θέση να κάνουμε μία πλήρη και απόλυτα ασφαλή χρήση όλων των μέσων PNR για να επιτύχουμε τους στόχους μας, αν δεν κάναμε χρήση ουσιαστικά όλων των παραμέτρων και χρησιμοποιούσαμε μόνο κάποια συγκεκριμένα μέσα ή εργαλεία στο πεδίο της ασφάλειας και της επιβολής του νόμου. Δεν πρόκειται λοιπόν για αυτή την πτυχή. Και που μπορεί να λειτουργήσει. Κατανοούν λοιπόν τα κράτη-μέλη ότι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι θα έλεγα μια λειτουργική προσέγγιση και θα πρέπει να αξιολογηθεί αντίστοιχα από τον εισηγητή τι μπορεί να γίνει. Έχετε κάποιες παρατηρήσεις κύριε Κέρκοπ να ολοκληρώσετε, να, να πείτε ολοκληρώνοντας. Θα ήθελα απλά να επαναρθώσω κάποιες παρανοήσεις που υπάρχουν πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, αυτό που προσπαθώ να κάνω, και εγώ είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τις ε, παρατηρήσεις που έγιναν και από τον συνάδελφο της Επιτροπής Μεταφορών, αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να δούμε, να προσεγγίσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να την θέσουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όσον αφορά τις ανταλλαγές πληροφοριών και δεδομένων στην Ευρώπη και να δούμε επίσης τι μπορεί να γίνει σε σχέση με άλλες συμφωνίες PNR και που εμπλεκόμαστε εμείς δραστήρια σε αυτές. Και μία αναφορά στην συμφωνία ΕΕ Αυστραλίας και πόσο θετική είναι και πόσο προσεκτικοί είμαστε και συνετοί σε αυτή τη συμφωνία για την προστασία ατόμων και προσωπικών δεδομένων τους. Να ληφθούν υπόψη όλες οι ανησυχίες που εξεφράστηκαν από τους συναδέλφους απόψε για τις προτάσεις που εγώ σκοπεύω να συντάξω και να υποβάλω στην ίδια την δική μου έκθεση. Αυτό είναι το εγχείρημα στο οποίο εμπλέκομαι. Είμαι ευγνώμων για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σίγουρα και ελπίζω ότι από αυτές τις συζητήσεις ίσως οι συνάδελφοι θα ξαναδούν πρώτα απ' όλα τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να ξαναδιαβάσουν πάλι τη Συμφωνία ΕΕ Αυστραλίας, να την ξαναδούν και πιστεύω ότι έχοντας πραγματογνωμοσύνη προσεγγίζοντας αυτό το θέμα μπορούμε να συνεργαστούμε για να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα. Διαφορετικά δεν χρειάζεται να γίνει αυτό και οποιαδήποτε συμφωνία με οποιαδήποτε άλλη χώρα θα μπορούσε να γίνεται εκτός αυτών των διαδικασιών. Αν όμως θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των πολιτών της με υπεύθυνο πνεύμα να εργαστεί. Πρέπει να συνεργαστούμε εμείς με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει σωστός έλεγχος και σωστός συντονισμός και τότε πρέπει να έχουμε, πιστεύω, συμφωνίες PNR που θα είναι λειτουργικές. Θέλω να ευχαριστήσω για το έργο της ε, τρέχουσας προεδρίας, της Πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτή τη συνεργασία που ήταν πολύ επικοδομητική φαίνεται σε ένα χρονικό πλαίσιο ότι δεν θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα αποκομίσουν, θα δρέψουν τους καρπούς τελικά από αυτή την προσπάθεια. Παρόλα υπάρχει μια πολύ θετική ανταπόκριση. Ακούσατε ότι υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές όσον αφορά Συμβούλιο και Επιτροπή, όσον αφορά κάποιες ε, συνιστώσεις. Θέλω να σας πω ότι άκουσα κάποια πολύ ενδιαφέροντα θέματα και παρατηρήσεις όσον αφορά κόστος και δαπάνες. Δεν δέχομαι συλλήβδιν όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι όπως προανέφερα για την ασφάλεια των πολιτών μας, το επίπεδο κόστους είναι πραγματικά πολύ χαμηλό για το τελικό όφελος προστασίας τους, ε, περί των ζωών των ανθρώπων αυτών, της ζωής τους. Πρέπει να μας ενδιαφέρει και να μεριμνήσουμε για την ασφάλειά τους, τη ζωή τους, αλλά και τα προσωπικά τους δικαιώματα, τα προσωπικά τους δεδομένα, την προσωπική τους ιδιωτική ζωή και το σεβασμό της. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε λοιπόν να προχωρήσουμε έτσι. Οι συνάδελφοι οι οποίοι ήταν, άσκησαν ιδιαίτερα επικρίσεις, ελπίζω ότι άσκησαν επικρίσεις επί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι επί των δικών μου προσεγγίσεων και προτάσεων. Θα ήθελα έτσι να προσεγγίσουμε το θέμα από κοινού επικοδομητικά. Θα κάνω ό,τι μπορώ να ενημερώνω τους σκιώδεις εισηγητές συναδέλφους και τον, τους συναδέλφους της Επιτροπής Μεταφορών και ελπίζω θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα στο τέλος τέλος. Ευχαριστώ. Ε, so much for today. Ε, and are... Αυτά για σήμερα στο συγκεκριμένο θέμα. Θα δούμε πώς θα γίνουν οι συζητήσεις στη συνέχεια. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν. Να σας δώσω κάποιες πληροφορίες. Θα υπάρξει ακρόαση της Επιτροπής μας για την εφαρμογή της χάρτας των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μετά από δύο χρόνια από την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Στις 23 Νοεμβρίου η επόμενή μας συνάντηση. Θα τα πούμε τότε.